Guten Μέρα, καλό απόγευμα κύριε και κύριοι. Ξεκινάμε με τη συνεδρίασή μα. Παρακαλώ καθίστε. Έχετε ενώπιον σα την ημερησία διάταξη. Και έχω τη μία αίτηση του κυρίου Μπουλόν, το σημείο 7, να το προτάξουμε και να γίνει σημείο υπαριθμών 4 για αύριο. Η κυρία Ράπτη έχει ζητήσει η γνωμοδότησή της να ψηφιστεί μετά το σημείο 19. Η κυρία Γκένς επίσης θέλει η δική της γνωμοδότηση η οποία είναι το 27 να προταχθεί του σημείου 24 και η συζήτηση για το φορέα του Τωρίνου Επαγγελματική εκπαίδευση, το σημείο 28 θα συζητηθεί μετά το σημείο 24, δηλαδή περίπου στις 5 το απόγευμα αύριο. Αν δεν έχετε λοιπόν άλλες αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Έχουμε στο σημείο 3, 2 μάλλον, πρακτικά της 24 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου και 26 27 Μαρτίου 2012 όσο δεν διατυπωθεί κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Τρία. Ανακοινώσει Πρόεδρου. Θα ήθελα να χαιρετήσω ένα νέο μέλος της Επιτροπής μας, πρόκειται για την από τη Ρουμανία, από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Καλώς ήλθατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, στην Επιτροπή μας. Επίσης θέλω να σας αναφέρω ότι έχουμε το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών μας. 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα έχουμε μια έκτακτη συζήτηση για την ε, γνωμοδότηση για τα κοινωνικά θέματα και για την ε, γνωμοδότηση επίσης του κ. Πόστελ σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία Προβλέπεται επίσης μια προσωρινή μερισσία διάταξη για την συνάντηση της 18 Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν όμως είναι υπερπλήρηση η ημερησία διάταξη, γι' αυτό θα ζητήσουμε μισή μέρα παραπάνω, το απόγευμα δηλαδή της 17 Σεπτεμβρίου. Θα σας αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις νέες ημερομηνίες. Και επιπλέον, στον φακελό σας θα βρείτε κάποια σημειώματα για την συνεδρίασή μας της 1ης Μαρτίου που συζητήσαμε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και το, η γραμματεία μας ανέλαβε να συντάξει ένα ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα αυτά για τη συζήτηση αυτή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Επιπλέον θέλω να σας υπενθυμίσω ότι διαδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και θέλω να χαιρετήσω και την έλευση της κυρίας Brody Commons στο προσωπικό της Γραμματείας της Επιτροπής Απασχόληση. Ερχόμαστε λοιπόν κατευθείαν στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης που γίνεται νέο σημείο 4 είναι η εντολή για το τριμερή διάλογο του προϋπολογισμού του 2013 με εισηγητή τον κύριο Φίλι Μπουλάου. Θα συζητήσουμε για τις τροπολογίες. Υπάρχουν ε, και τροπολογίες συμβιβασμού. Όλα αυτά θα ψηφιστούν, όλες αυτές οι τροπολογίες θα ψηφιστούν αύριο το πρωί, αλλά θα ήθελα να δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να τοποποιήσετε την ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν θέλετε να επανέλθω για τον προπολογισμό 2013, γιατί πριν από λίγες ημέρες το παρουσιάσαμε ε, στην Επιτροπή ε, απασχόλησης. Ε, όλο και περισσότερο αναφέρονται τα ζητήματα της απασχόλησης. Έχουμε, το θέση, έχουμε τονίσει ιδιαίτερα ε, τα προγράμματα Progress, ΕΡΕΣ, τα προγράμματα της απασχόλησης, την απασχόληση των νέων ειδικότερα και την στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αυτές που υπόσχονται τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους. Για τον προϋπολογισμό του 2013 έχουν κατατεθεί 29 τροπολογίες και από τους σκιώδους συζητητές των άλλων ομάδων. Τους ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις συμβιβαστικέ και όχι πέντε. Ε, έχουν γίνει αποδεκτές από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Ε, ο συμβιβασμός ΣΥ αποσύρθηκε από την ΚΟΕ και η κυρία Γκένς αρνήθηκε Οπότε θα ψηφίσουμε τις 10 και τις 11 που είναι συμβατές και θέλει ε, η κυρία Γκέντς να προσθεθεί μία φράση που υπήρχε στο συμβιβασμό C, έναν ουδέτερο προϋπολογισμό που δεν έχει επίδραση στην κοινωνική προστασία. Εγώ ως εισηγητής θέλω βεβαίως να υποστηρίξω τις τέσσερις συμβιβαστικέ τροπολογίες, ε, επίσης την τροπολογία 16, 9, 24, 26, 27 των σοσιαλιστών και 18 των πρασίνων αλλά θα ήθελα να καταψηφίσουμε κάποιες τροπολογίες, την υπαριθμόν 3 για παράδειγμα, του κυρίου Μπροκ ε, που αναφέρεται στην πραγματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση των νέων. Επίσης, τη 17 ε, του ιδίου συναδέλφου που προτείνει μία προσαρμογή της ε, πολιτικής ε, για την απασχόληση των νέων και ε, προτείνω να τη συμπεριλάβουμε να ψηφίσουμε αντί για την 17 την 19. Προτείνουμε επίσης να καταψηφιστεί η τροπολογία των μη εγγεγραμμένων γιατί μου φαίνεται ότι αυτό που προτείνει δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οι τροπολογίε 22, 23, 25 ε, τις οποίες προτείνω να καταψηφίσουμε επίση, γιατί είτε είναι ασύμβατες ε, ε, με την ε, νέα δημοσιονομική γραμμή για την προστασία της επισφαλούς απασχόλησης, κυρίως γιατί η τροπολογία 22 δεν είναι αρκετά ακριβής. Αυτή είναι η προσέγγιση που προτείνω εγώ να ακολουθήσει η Επιτροπή μας ε, για την γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό 2013. Ευχαριστώ πολύ. Als nächstes der Kollegin Darden. Ο κύριος Νταρντέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια να πω μόνο ότι χαίρομαι για τη θέση του εισηγητή τόσο στην πρόταση που αφορά τις ψηφοφορίες, όσο και στις προτινόμενες συμβιβαστικές ε, λύσεις όπου ενσωματώνονται στοιχεία σημαντικά όπως η ανάγκη κινητοποίησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ώστε να ε, επιτύχουμε τους στόχους ε, της στρατηγικής 2020, την αξιοποίηση του ΦΕΜ επίσης, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και διάφορα θέματα για τα οποία συμφωνούμε και άρα θα στηρίξουμε και εμείς τις συμβιβαστικές τροπολογίες που αναφέρθηκαν. Then, Κυρία Ζουμπέρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τις τροπολογίες μας. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Εμείς θεωρούμε ότι ιδίως σε μια χρονική στιγμή κρίσης και διάβρωσης πολλών δικαιωμάτων, ιδίως εργασιακών δικαιωμάτων που είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των κονδυλίων που ενισχύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σαν στόχο να προωθήσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς κυρίως στις χώρες οι οποίες έχουν φυγεί περισσότερο. Έχουμε λοιπόν καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες που μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι φιλόδοξες ή ότι, ότι εκφεύγουν, μέσα, εκφεύγουν από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά πιστεύουμε νομίζουμε ότι, ότι παρά το γεγονός ότι δεν συνάπτονται όλα αυτά τα στοιχεία του παζλ με ένα σαφή τρόπο, πιστεύουμε ότι κάθε επιτροπή έχει το καθήκον να πράξει τα αναγκαία στο δικό της τομέα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να καθορίσουμε από την πλευρά της Επιτροπής μας την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι το να μην μπούμε τίποτα σε σχέση με την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων θα ήταν κάτι σε αντίφαση με τη γενική μας στάση. Και νομίζω γι' αυτό το λόγο ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική στάση υπέρ μιας τέτοιας αύξησης. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο. Ξαναδίνω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους κατέθεσαν τροπολογίες και όσους ε, αποδέχθηκαν τις συμβιβαστικές τροπολογίες τους. Ευχαριστώ επίσης. Αυτή, σε αυτή τη γνωμοδότηση είναι σημαντικό να μην αρκεστούμε στη διευθέτηση των ε, τελευταίων δαπανών ενός ε, ε, πολιετούς ε, δημοσιονομικού ε, πλαίσιου, γιατί είναι πολύ σημαντικό στη γνωμοδότηση αυτή να τονίσουμε μια δυναμική η οποία πρέπει να συνάδει με την πραγματικότητα, με την απασχόληση κυρίως των νέων. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει λοιπόν αυτό το σημείο και περνάμε στο προηγούμενο τέταρτο σημείο πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας στις 7 Απριλίου συζητήσαμε το θέμα αυτό. Έχουμε τώρα 46 τροπολογίες και 7 τροπολογίες συμβιβασμού και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Χουισμένοβα. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο σκιώδη εισηγητές για την καλή του δουλειά, τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητά τους. Όσον αφορά το σχέδιο πρότασης, υποβλήθηκαν 46 τροπολογίες και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό βελτιώνουν την ποιότητα της γνωμοδότησης. Μετά από βαθιές συζητήσεις, Φτάσαμε σε έξι συμβιβαστικές τροπολογίες. Και διάφορες τροπολογίες που υποβλήθηκαν βασικά από δύο πολιτικές ομάδες. Εγώ βρίσκω πως η συμπερίληψη του κειμένου για την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και της, ε, του αποκλεισμού πολύ σημαντικές καθώς και τις διατυπώσεις που αφορούν την πρόσβαση στην ε, υγειονομική περίθεψη όταν πρόκειται για απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές που υποφέρουν από δημογραφικές αλλαγές. Συμβιβαστική F ε, στηρίζεται πολύ σίγμα ΚΑΤΑΦ στηρίζεται πολύ από τις πολιτικές ομάδες και ε, προκύπτει από τη βαθιά ανάλυση και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών των διαφόρων εδαφών, ιδιαίτερα αυτών που υποφέρουν από την απασχόληση, από την ε, ανεργία και την φτώχεια, καθώς πράγματα που οδηγούν στις διακρίσεις και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Είμαι τη άποψη ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η εδαφική προσέγγιση και θα πρέπει να είναι ένα φιλόδοξο ε, μηχανισμό για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εξέβρεση νέων βιώσιμων θέσεων απασχόληση. Για το στόχο αυτό χρειαζόμαστε προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση, για την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων, καθώ και την ενθάρρυνση τη επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται εξίσου η ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώ και ε, μαθήματα κατάρτισης για τους ε, εργαζόμενους γιατί οι θεσμικές δυνατότητες των διαφόρων επιπέδων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την επιτυχία της εδαφικής προσέγγισης και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Είμαι ευτυχής που η θέση μου έχει βρει συνένεση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στη βελτίωση του κειμένου προς αυτή την κατεύθυνση. Η συμβιβαστική G σχετίζεται με την αρχή της εταιρικής σχέσης και στηρίζεται ευρύτερα από τις πολιτικές ομάδες. Συμμερίζομαι την σημασία για την καλή σχέση μεταξύ της ε, πολιτικής συνοχής και των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα του κοινωνικού τομέα. Ε, επίσης, ε, είναι συμπληρωματικότητα των μέτρων που χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα και σε διάφορα επίπεδα όπως για την παιδεία και την υγεία. Οι τροπολογίες τις οποίες όμως δεν στηρίζουν είναι πολύ λίγες και αυτό δεν οφείλεται στο ότι απορρίπτω τι ιδέες που περιλαμβάνουν, που εμπεριέχουν, αλλά λόγω των ε, συζητήσεων που είχαμε σε διάφορα βήματα. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για να μπορούμε να λαμβάνουμε σωστά τις αποφάσεις μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για τη συνεργασία της και επίσης και σκιώδης συζητήσεις στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να συμπεριληφθεί αυτή η γνωμοδότηση στην τελική εκδοχή της έκθεσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ από τους πράσινους ως η εισηγήτρια κυρία Σρέντερ. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία που είχαμε μαζί της έχουμε βρει σημεία ε, σύγκλησης με την εισηγήτρια. Θέλω να τονίσω ότι αυτό που για μας είναι το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι μέσα από τις τροπολογίες και φυσικά μέσα από το κείμενο που έχει ήδη διατυπώσει η ίδια η να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα του πώς ή με ποιους τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την έννοια της κοινωνικής κατανάλωσης. Υπάρχει το πρόβλημα του ΑΕΠ που ξέρουμε ότι ως ε, μέτρο μέτρησης δεν είναι επαρκές. Χρειαζόμαστε να έχουμε κοινωνικά κριτήρια για να περιγράψουμε αυτή την έννοια της κοινωνικής κατανάλωσης των κοινωνικών αγαθών, ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Ευρώπης, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κατατεθούν οι αντίστοιχε τροπολογίε και να επιτύχουμε τι κατάλληλε συμβαστικέ λύσει, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη σε αυτή την έκθεση και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε μια καλή προοπτική για την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάρντεν και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και εμείς υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες και συγκεκριμένα όσον αφορά τη σημασία της ε, κατάρτασης των τοπικών και περιφερειακών αρχών ε, ε, την ε, χρήση ε, των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου, όπως επίσης και τη χρήση των διαδοτικών ταμείων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την απαραίτητη κάλυψη από τα διαδοτικά ταμεία του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και Ελπίζουμε να είναι υπέρ των τροπολογιών αυτών ή τουλάχιστον να καλύπτονται από τις συμβιβαστικές της ε, εισηγήτριας. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση, ε, τις οποίες υποστηρίζει δική μας ομάδα και η ομάδα των Πρασίνων ε, και όχι από όλε τις ομάδες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα περάσουν. Θα δούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας να θα γίνει αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, συνεργασία της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότηση της κυρίας Μενόβα και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που ελέγχθηκε από τους άλλους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή εργασία και προσδοκώ ότι το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία αύριο. Μόνο δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να προσφέρω στη συζήτηση. Νομίζω υπάρχουν μερικά σημαντικά στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω και στους συναδέλφους. Εμείς επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής μας προκύπτει από την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η συνοχή σημαίνει γεωγραφική συνοχή, οικονομική συνοχή, κοινωνική συνοχή. Πιστεύω όμως ότι μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση και οι αναφορές που κάνουμε σε μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση παραμένουν μονάχα συμβολικού χαρακτήρα, ότι δεν υλοποιούνται με τις ενέργειές μας και τις πράξεις μας στη συνέχεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα αυτό μετά από το 2013. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα θέματα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ξεπεράσει το επίπεδο συνθημάτων και μόνο και θα πρέπει να αποδώσουμε την πρέπουσα σημασία στις πολιτικές απασχόλησης μέσα στο στον πολιτικό χώρο της συνοχής και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τις ποικίλε και διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι περιφέρειες της Ευρώπης. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η εξής. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία έχει σημασία λέγω, η Επιτροπή Απασχόλησης να υποστηρίξει τις τροπολογίες οι οποίες θα έκαναν το όλο σύστημα να είναι πιο ευέλικτο γιατί με ένα τέτοιο πιο εύκαμπτο σύστημα θα ήταν πιο εύκολο για τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης να εφαρμόσουν τα ενωσιακά σχέδια. Ελπίζω ότι θα ψηφίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση αύριο. Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος. Ξαναδίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Χιουισμένοβα, στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μία ακόμη φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές και θα ήθελα να επισημάνω ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα, γιατί συνεισφέρουν στην ποιότητα του κειμένου και πιστεύω ότι ελπίζω στο μέλλον ε, να έχουμε και πάλι τόσο καλή συνεργασία προκειμένου να, είναι, να προκύψει ένα πολύ καλό ενοποιημένο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα γίνει αύριο η ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Περνάω στο σημείο 5. Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονία. Και εδώ η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Σιλβάνα Ράπτη. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά την έκθεση Κούκαν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων <clears throat> και έχουμε τώρα 50 περίπου τροπολογίες. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγητρία την κυρία ράπη, για να συζητήσει για τις τροπολογίε αυτές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω μετρήσει γύρω στις 40 τροπολογίες ε, και έχω καταλήξει σε 10 συμβιβαστικές. Στις ε, συμβιβαστικές που έκανα προσπάθησα όσο μπορούσα ε, να κάνω το κείμενο συνολικά της γνωμοδότησης ε, περισσότερο σαφές και με όσο το δυνατόν καλύτερη δομή. Ε, έκανα και κάποιες αλλαγές μετά από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι Σκιώδης και τους ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους και οι πολιτικές ομάδες, ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έχει σημασία αυτό για μένα θέλω να σας πω ότι ε, ε, επιτρέψτε μου να έχω την εντύπωση ότι έχουμε διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές προτάσεις για τους γείτονές μας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι το κείμενο της πρότασης του κανονισμού χωρίς αυτή τη γνωμοδότηση την οποία ξεκίνησα εγώ αλλά εμπλούτησαν στην πορεία οι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες, δεν θα υπήρχε σχεδόν καμία αναφορά σε ζητήματα απασχόλησης, ε, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών δικαιωμάτων. Άρα θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει συλλογικά και όχι μόνο από μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρία πράγματα θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει. Το πρώτο είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων με ειδική φροντίδα και μέρημνα για τις ευάλωτες ομάδες. Το δεύτερο είναι να υπάρχει αναφορά και συγκεκριμένες κατά το δυνατόν προτάσεις για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ενσωμάτωση. Και το τρίτο είναι ότι προβλέπουμε πράγματα, σημεία που έχουν να κάνουν με τη στήριξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Ε, πιο ειδικά ζητάμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για θέματα κοινωνικής προστασίας. Ζητάμε να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Ζητάμε να βελτιωθούν οι πολιτικές απασχόλησης και σε αυτές να περιλαμβάνονται και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ζητάμε να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και βεβαίως να αντιμετωπίζονται οι καταχρήσεις στην αγορά εργασίας. Ζητάμε να επικυρωθούν οι σημαντικότερες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ζητάμε να ελέγχεται η κυκλική κινητικότητα. Ζητάμε επίσης θεσμούς που θα διευκολύνουν το να συναντώνται η ζήτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων και των εργοδοτών με την προσφορά από, τις, από τους εργαζόμενους σε κάθε περιοχή ανάλογα με τις δεξιότητες που διαθέτει κάθε περιοχή. Επίσης, ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρέωση διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών πριν από την θέσπιση νόμων. Και βεβαίως θέλουμε να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Τελειώνοντας, ε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά, σημαντικό, ε, εξαιρετικά σημαντικός ο περιοδικός έλεγχος για συμμόρφωση των γειτονικών χωρών με αυτά τα οποία ζητά, ε, ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον έλεγχο αυτό πρέπει να βλέπουμε κατά πόσον γίνεται πρόοδος σε σχέση με αυτά που προτείνουμε εμείς μέσα από αυτή τη γνωμοδότηση. Εδώ βάζω τελεία. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τους σκιώδεις συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες και βεβαίως τη γραμματεία και τους συνεργάτες μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. E ο έχει από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το πολύ καλό έργο της. και για τις ε, τροπολογίες της που βελτιώνουν αυτή την έκθεση. Είναι σημαντικό <clears throat> να έχουμε στην πολιτική γειτονία μας ένα, γειτονίας μας ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί να παρακολουθήσει τη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον περιγυρό μας και να έχουμε και τους κατάλληλους, δίκ, τους δείκτες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την εποπτεία της δαπάνης αυτών των κονδυλίων. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα του ΕΛΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτή τη γνωμοδότηση εκτός από δύο <clears throat> τροπολογίες, τη συμβιβαστική H λατινικό. Πιστεύουμε ότι εκεί το κείμενο προχωράει υπερβολικά όταν μιλάμε για την πρόθεση της κινητικότητας των πολιτών και την πρόθεση των επαφών μεταξύ αυτών. Στη συμβαστική αυτή όμως τροπολογία Ο κύκλος αυτός κινητικότητας, η κυκλική κινητικότητα είναι μια διατύπωση που δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Ίσως υπάρχει κάποια ασάφεια στην διατύπωση και η ασάφεια αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Γι' αυτό δεν μου αρέσει αυτή η συμβαστική τροπολογία H. Και η διατύπωση εδώ για τα κονδύλια που απαιτούνται νομίζω ότι κάπως ξεπερνά και ως μέσα από τις των συναδέλφων. Έχουμε πει στη συμβαστική τροπολογία C και αυτή έχει να κάνει ως με, με σημαντικά θέματα. Είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμπερίληψη και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βεβαίως, είναι σημαντικά αυτά. Όταν λέμε όμως ότι αυτή πρέπει να είναι οι στόχοι να είναι εγκάρσιοι στόχοι σε όλες τις δράσεις που υπόκεινται σε αυτόν τον κανονισμό και αυτό νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό. Εγώ θα έλεγα ότι η ισότητα των φύλων, η μη διακρίσεις ως αρχή, η κοινωνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να λειτουργήσουν έτσι αλλά η κοινωνική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των εργαζομένων ότι θα πρέπει να είναι πάντα μόνιμες εγκάσεις αρχές σε όλες μας τις δράσεις δεν συμφωνώ. Γι' αυτό εμείς είμαστε εναντίον στο δικό μας κατάλογο ψηφοφορίας. Κατά τα άλλα όμως θεωρώ ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι εξισορροπημένα διατυπωμένη και νομίζω ότι θα δώσουμε την πρέπουσα υποστήριξη σε αυτήν αύριο το πρωί στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο από την Κομισιόν που θα ήθελε να λάβει θέση για, αυτό το, για αυτή την γνωμοδότηση. Υπάρχει κάποιο αρμόδιος. Όχι. Ξαναδίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Ράπτη το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ε, δεν περίμενα να πάρω το λόγο τόσο γρήγορα. Άλλη σκιώδης ε, να νιώθω, να αισθάνομαι ευχαριστημένη δηλαδή. Μου έχετε πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Καλό είναι αυτό λέω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Σάρη για μια ακόμη φορά για τις παρατηρήσεις της ε, και να πω το εξής, σε σχέση με την κυκλική κινητικότητα, αν μπορώ να το πω με απλά λόγια, είναι το εξής. Καταρτίζουμε, εκπαιδεύουμε προσωπικό από τις γειτονικές χώρες, δίνουμε τεχνογνωσία, αλλά όταν το προσωπικό αυτό πάρει την τεχνογνωσία και τις γνώσεις, θέλουμε να γυρίσει πίσω στη χώρα, ώστε τη γνώση, την τεχνογνωσία που πήρε να τη χρησιμοποιήσει σε αυτές τις χώρες και στους λαούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα να φεύγουν κορίτσια και αγόρια, πρικισμένα μυαλά, να έρχονται α, στην, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παίρνουν γνώσεις, να παίρνουν τεχνογνωσία και μετά να φεύγουν από τις γειτονικές μας χώρες και να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ουσιαστικά συμβάλλουμε χωρίς να το θέλουμε στην, ε, πώς το λέμε, έχουμε έναν όρο που δεν τον θυμάμαι τώρα, στο να παίρνουμε εγκεφάλους, ε, brain train, με βοηθάει η ναι, Αντιγόνη, brain train brain train. Συμβάλλουμε χωρίς να το θέλουμε σε αυτό. Αυτό είναι η αίσθηση, αυτό που λέμε κυκλική κινητικότητα. Να παίρνουν τη γνώση, να παίρνουν την τεχνογνωσία και να γυρίζουν πίσω στις χώρες τους να τις αξιοποιούν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό που λέει η Σάρη ότι ε, προχωράμε πολύ και στην ε, ε compromise ε, H και στην συμβιβαστική σε. θέλω να το δω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διατηρηθεί η συμβιβαστική, αλλά έχω στο μυαλό μου ότι μερικές φορές ίσως να είναι καλύτερα να πηγαίνουμε λίγο πιο μπροστά, προσπαθώντας να σώσουμε ε, πράγματα που έτσι κι αλλιώς κινδυνεύουν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σαν Σιλβάνα, αλλά και ως πολιτική ομάδα, ως σοσιαλιστές, έχουμε ε, αυτή την πολύ μεγάλη ευαισθησία που και, το EPP έχει σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, γι' αυτό ακριβώς έχω πολύ μεγάλη α, έγνοια. Γι' αυτό λαμβάνω πολύ μεγάλη ε, μέρημνα και φροντίδα. Ε, να το δούμε και ε, να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και την ε, Σάρη και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και σας κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί, θα ψηφιστεί αύριο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιούλιο. Έρχομαι στο σημείο 6, Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017. Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο συνάδελφος Σανταμ Κούσα από το ΕΛΚ. Υπάρχουν 40 τροπολογίες και υπάρχουν και οι προτάσεις συμβιβασμού που έχουν κατατεθεί επίσης. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Κούσα. Δεν μπορεί να είναι παρόν ο κύριος Κούσα εδώ σήμερα και θα συνεχίσω εγώ και θα σας τα πω και στα Ουγγρικά. Τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Επασχόλησης Συζητήσαμε τις τροπολογίες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017 και σε επικίνδυνη ευκαιρία είχα πει ότι ε, μεταξύ των σημαντικών στόχων του προγράμματος που διέπει τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, υπήρχε και η ανάγκη συλλογή στοιχείων ε, πιο περιστατωμένων και σε περισσότερα επίπεδα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να μιλάμε για τις ίδιες έννοιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τότε μιλήσαμε για την ανάγκη πρόσβασης στα στοιχεία και είχαμε πει ότι οι ερμοδιότητες, των, τα καθήκοντα μάλλον των κροτών μελών πρέπει να είναι αντίστοιχα με τα καθήκοντα και τις προκλήσεις και άρα ήταν σημαντικό να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, κυρίως επειδή οι ειδικοί και οι αναλυτές είναι αυτοί που εκφράζονται με τις ίδιες έννοιες. Έγιναν λοιπόν ένα σωρό προτάσεις τροπολογίε ανάμεσα στην ε, συνεδρίασή μας, ε, την προηγούμενη και τη σημερινή και στις 23 του μηνός στο Στρασβούργο καταφέραμε να εκπονήσουμε 8 συμβιβαστικέ τροπολογίες που συμπεριλαμβάνουν ε, καμιά τριανταριά τροπολογίες. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες τις οποίες δεν υποστηρίζω, γύρω στο 33%, αλλά πάντως μπορέσαμε να δεχτούμε τα δυο τρίτα των τροπολογιών τροπολογιών. Αυτές οι τροπολογίες τις οποίες δεν στηρίζω αφορούσαν τεχνικές στατιστικές επιτυχίες που θα μπορούσαν περαιτέρω να περιπλέξουν τα πράγματα ή να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή εξέλιξη των προγραμμάτων. Επειδή εδώ μιλάμε για κανόνες οι οποίοι διέπουν, μάλλον ορίζονται, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και μετά υπάρχει μια σειρά θεμάτων όπου δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει πάντοτε να εντάσσονται όλα αυτά στον τρόπο εργασίας της Κομισιόν. Αυτά και ευχαριστώ. Euh, ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου και μετά στην κυρία Ντελή για τους πράσινους. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, κάναμε συνεδρία των Σκιωδών στο Στρασβούργο στις 23 Μαΐου, που ήταν πολύ καλό, διότι διαβάσαμε όλες τις τροπολογίες και τις συζητήσαμε. Και είχαμε συμβιβαστικές οκτώ τις οποίες θα δεχτούμε. Η ομάδα των σοσιαλιστών υπέβαλε διάφορες τροπολογίες, ορισμένε εξ αυτών δεν έγιναν δεκτέ από τον κύριο Κόσε και για να σας πω την αλήθεια πιστεύω 8 από αυτέ αναφέρονταν στην ανάγκη για υψηλή ποιότητα στατιστική, ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να σχεδιάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές που είναι μάλιστα ένα από του κυρίω στόχου του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματο και ε, είναι και σύμμορφο προς τους ευρύτερους στόχους της Ένωσης. Ε, εγώ πιστεύω πως οι οχτώ αυτές τροπολογίες που τονίζουν την υψηλή ποιότητα των ε, στατιστικών θα γίνουν δεκτές, θα ψηφιστούν από κοινό αύριο και ελπίζω πως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα τις υποστηρίξουν. Όσον αφορά το στόχο των σοσιαλιστών είναι να έχουμε και να μπορούμε να διαδώσουμε και καλή ποιότητα στατιστικές που χρειάζονται οπωσδήποτε σε μια φάση οικονομική κρίση, γιατί οι αποφάσει θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση ε, και συγκρίσιμε στατιστικές. Έχουμε επίση καταθέσει κάποιε προφορικέ τροπολογίε ω ομάδα και σε μια από αυτές τονίζουμε την ανάγκη το κονδύλι για το πρόγραμμα να καταναμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν οι απαραίτητες δαπάνες για τη βελτίωση των διαδικασιών και δυνατότητε δυνατότητες εκπόνησης ε, κατάρτισης ε, ψηλής ποιότητας στατιστικών σε εθνικό επίπεδο. Εν γέννη, η έκθεση αυτή θα υπερψηφιστεί νομίζω από την πλειοψηφία αύριο για την καλή έκθεση και οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί την βελτίωσαν ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κυρία Ντελή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του, θα ήθελα να επιμείνω σε τρία σημεία που αναφέρω και στις τροπολογίες μου, για τις οποίες θα ήθελα μάλιστα να ζητήσω και την υποστήριξή σας. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τις πολιτικές μας μέσω από ένα πρίσμα ε, χρηματοοικονομικό και μακροοικονομικό. Η κρίση δεν πρέπει να μας κάνει να μην βλέπουμε τα σημαντικά ε, πράγματα που είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες, η οργάνωση της κοινωνίας μας. Ε, ε, αυτή η κοινωνία δημιουργεί την οικονομία και όχι το αντίστροφο. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να πιέσουμε για την ενίσχυση της ποιότητας και της ποικιλία των κοινωνικών δικτών και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να δώσουμε τις βάσεις για μια πραγματική κοινωνική πτυχή και της παγκοσμιοποίησης αλλά και των οικονομικών πολιτικών μας. Συμφωνώ επίσης με το να τονίσουμε την αποτελεσματικότητα ε, του κόστους ε, ε, της προσπάθειας που γίνεται στο πλαίσιο της, του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος. Αλλά προσοχή, θα ήταν αντιπαραγωγική ήλιτο η λιτότητα, ενώ όλοι μιλούν για την, το, το πόσο προστιθέμενη αξία έχει η στατιστική παραγωγή, ο συντονισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι ότι οι στατιστικές πρέπει να έχουμε και στατιστικές για τη στέγαση. Είναι μια προτεραιότητα των συμπολιτών μας των Ευρωπαίων και ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση και αυτό πραγματικά ένα μια πρόκληση με κύρια πρόκληση του αστέγους ε, που είναι άνθρωποι που πλήττονται ιδιαίτερα από ε, την φτώχεια και πρέπει εμείς ως εκλεγμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτό το θλιβερό φαινόμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριος Μπενιάμ. Ναι, ναι, συγγνώμη, δεν είχα τα ακουστικά μου και δεν σας άκουσα στην αρχή. Δεν έχω να πω πολλά, γιατί ουσιαστικά συμφωνούμε με την εισηγήτρια και το τόνισα και στην αρχή. Υπήρξαν μονάχα ορισμένε γλωσσικές διευκρινήσεις που θέλησαμε να επισημάνουμε και συμφωνούμε σε όλα τα θέματα, εκτός από το θέμα των στατιστικών υψηλής ποιότητας. Για μένα είναι ένα πρόβλημα νομικού ορισμού, αλλά η συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και οι συμβαστικές τροπολογίες που πρόκυψαν νομίζω ότι αντανακλούν μία συνένεση και επίσης η προφορική τροπολογία της κυρίας Παπαδοπούλου η οποία μας βρήκε σύμφωνος. και πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ καλή διαδικασία επίτευξης συνένεσης και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν ο οποίος ενδεχομένως θα ήθελε να λάβει το λόγο. Εντάξει, δεν ζητεί κανείς το λόγο. Θα ξαναδώσω ο κύριος ε, Οντί, ο, ο Ρή μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συγγήτρια έπρεπε να πάει σε μια άλλη επιτροπή. Απλώς για να συνοψίσω αυτή τη συζήτηση, εγώ έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Πιστεύω το κείμενο το τελικό στο οποίο καταλήξαμε είναι γενικά αποδεκτό. και ούτε η γνωμοδότηση ούτε η έκθεση επί της ουσίας θα αντιμετωπίσουν και θα επιλύσουν το γνωστό πρόβλημα ότι τα 28 κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά στατιστικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν κάνει εύκολο να έχουμε συγκρισιμότητα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά νομίζω ότι ο κ. Κώσα και οι συναδελφοί του έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά και εξ ονοματός του θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συζητητές για τη συνεργασία τους και ελπίζω ότι θα περάσουμε μεγάλη πλειοψηφία η γνωμοδότηση αυτή αύριο. Ωραία. Αύριο θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση του κύριου Κούσα. Περνάμε στο σημείο 14 της ημέρησιας διαταξής μας. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, εγώ λέω άλλαντάλλον σήμερα. Περνάμε στο σημείο 8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ψηφίζουμε την γνωμοδότησή μα υπομορφή επιστολή για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι ένα κείμενο γενική χρειά γιατί αφορά την αίτηση τεχνικής αρρωγής που έχει παρουσιαστεί από την Κομισιόν. Εγώ δεν έχω λάβει καμία τροπολογία για το κείμενο αυτό της επιστολής. Σας προτείνω λοιπόν να την θέσουμε σε ψηφοφορία. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή η ψηφοφορία. Έχετε όλοι κάρτες. Εγώ όχι, αλλά θα ψηφίσω υπέρ όπως φαντάζεστε. Ανασπάσατε λοιπόν τα σκάρτα σας και άρχεται η ψηφοφορία. Ναι. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρασε ψηφοφορίας. Ναι, ναι, Όχι, δεν έκλεισε η ψηφοφορία, είναι ανοιχτή ακόμα. υπάρχει ένα, ένας βουλευτής που δεν έχει ψηφίσει. Περιμένουμε, περιμένουμε. Ωραία, κλείνω λοιπόν την ψηφοφορία. 32 ψήφισαν, 30 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Και στο σημείο 9 θα ψηφίσουμε την επιστολή η οποία αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση με συγκεκριμένα στην αίτηση της ε, Κομμουνιδάδ Βαλενθιάνα για τα θέματα υπόδηση. Δεν έχουμε και εδώ τροπολογία. Άρχεται και εδώ η ψηφοφορία, αλλά ηλεκτρονικά όπως πάντα. Εάν ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. 35 ψήφισαν, 32, 33 υπέρ, μία ψήφος κατά. Γίνεται δεκτή λοιπόν με ευρύτατη πλειοψηφία αυτή η επιστολή. Αυτά ήταν με τη σύντομη αυτή σειρά ψηφοφοριών. Αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερες, αλλά διακόπτω μια στιγμή τη συνεδρίαση για να ανακατανύμουμε τα προεδρικά εδόλια και να υποδεχθούμε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Συνδικάτων, την κυρία Μπεναντέ Σεγόν. de, reprendre nos travaux. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να καθίσετε για να ξαναρχίσουμε. Et j'ai euh, Με πολύ χαρά και με, είναι μεγάλη μου τιμή που πρώτη φορά θα είναι εδώ ε, από τότε που εξελέγει εδώ και ένα χρόνο Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκής Νομοσπονδία Συνδικάτων, η κυρία Μπερναντέτ Σεγκόλ. Μπορεί κάποιοι εξημών ε, να την έχουν συναντήσει. Ε, λόγω των συζητήσεων που γίνονται και στη δική μας Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη όμως η συνάντησή μας ε, για να γίνει μια γενική συζήτηση γύρω από τις προτάσεις ε, ε, από πλευράς του Επιτρόπου μας για το πακέτο της απασχόλησης, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια συνολική θεώρηση για τα ζητήματα αυτά, να εισαγάγουμε νέα σημεία στη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξισορροπήσουμε κάποια στοιχεία στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής ε, του Σώματος των Επιτρόπων ε, για την πτυχή της προσφοράς της πρότασης. Με όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Γενική Γραμματέα για μια μικρή παρουσίαση και θα έχετε ούτως ή άλλως στη συνέχεια τη δυνατότητα να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά τη διαδικασία. Αν μπορείτε εντός 15 λεπτών ε, να ολοκληρώσετε την παρουσίασή σας θα ήταν τέλεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Περβόνς. Ε, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που είμαι εδώ σήμερα να μιλήσω ε, για αυτό που ε, για την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, αποτελεί, όπως θα φαντάζεστε, το πρώτο σημείο των ανησυχιών μας, το ζήτημα της απασχόλησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ορισμένες χώρες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δραματική και δεν υπερβάλλω όταν χρησιμοποιώ αυτό ε, τον όρο. Και πρόκειται για μια κατάσταση που θέτει ένα αμφιβόλο την αξιοπιστία της ε, ευρωπαϊκής πορείας και την εμπιστοσύνη που ε, οι εργαζόμενοι και οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν στην όλη αυτή διαδικασία. Είναι λοιπόν σαφές ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να χαιρετήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει ένα πακέτο απασχόλησης και να ε, και την απόφαση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξαναθέσει στο επίκεντρο των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα της απασχόλησης. Στην παρέμβασή μου που θα προσπαθήσω να την ολοκληρώσω σε 15 λεπτά, θα προσπαθήσω να σας πω πού βλέπουμε τα θετικά ε, στοιχεία, αλλά και που βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβληματικά σημεία στο πακέτο αυτό απασχόλησης. Πρώτα απ' όλα για τα προβληματικά σημεία θα έλεγα ότι έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ε, σε σχέση με τη δυνατότητα του πακέτου αυτού να είναι αποτελεσματικό ε, αν λαμβάνει η χώρα εκ παραλίλου με τα ε, μέτρα λιτότητας που επίσης αποφασίζονται σήμερα αν δεν ε, φρενάρουμε λιγάκι, αν δεν υπάρχει μία πάυση για κάποιους μήνες ε, στα μέτρα αυτά, τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται ε, στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει ανάπτυξη που θα ευνοήσει την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας λοιπόν αυτό το θέμα ε, της συνέχισης ε, των μέτρων λιτότητας ε, και παράλληλα η ε, ύπαρξη μέτρων για την απασχόληση ε, δεν μπορεί να συμβαίνει, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τα δύο παράλληλα. Αυτό επίσης ε, που μας θλίβει στο πακέτο αυτό για την απασχόληση είναι ότι συνεχίζουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να επικεντρωνόμαστε στα διαρθρωτικά μέτρα. για την ε, ανάκαμψη της, ε, ε, της απασχόλησης. Όπως είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα δεν είναι μόνο η αύξηση της προσφοράς, αλλά να δούμε και το θέμα, να δούμε το θέμα της ζήτησης μάλλον. Από εκεί να αρχίσουμε. όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαρθρωτικά θέματα έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε μια λέξη που πολλά χρόνια την ακούμε, το θέμα της ε, ευέλικτης ασφάλειας, και παρά το γεγονός ότι έχει επιτύχει στις βόρειες χώρες, ε, στις σκανδιναβικές χώρες, ε, έχει συλληφθεί και εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες μέλη ως έννοια που επιτρέπει την πρόσληψη αλλά και την απόλυση ε, εργαζομένων και λιγότερος ε, προσπάθεια ε, μείωση της προστασίας που υπάρχει στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για τους εργαζομένους. Το θέμα αυτό λοιπόν της ευέλικτης ασφάλειας ε, ήταν ένα ζήτημα που είχε θεωρηθεί θετικό όταν ε, αφορούσε τις, τις ενεργούς πολιτικές ε, της απασχόλησης, όμως όταν εφαρμοζόταν στις διάφορες χώρες μέλη, τα πράγματα, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Ξέρουμε τι έγινε σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο, τις κοινωνικές σχέσεις σε συγκεκριμένες χώρες όπως για παράδειγμα παράδειγμα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Κάτι το οποίο παρεμποδίζει βέβαια ε, η έννοια αυτή ε, να θεωρείται θετική. Όσον αφορά τώρα το ε, ζήτημα της υποστήριξης της ενίσχυσης της απασχόλησης, της ε, παραγωγής ε, θέσεων απασχόλησης ε, και της ενίσχυσης κυρίως των προσλήψεων, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο, υπάρχει μία απόχρωση που υπονοεί ότι πρέπει να γίνει, να, δούμε τα ενδεχόμενα, τον ενδεχόμενο στρεβλό αντίκτυπο που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, δηλαδή το να απολύουν οι, εργα... οι εργοδότες κάποιους ε, ε, εργαζομένους για να τους επαναπροσλάβουν ε, προκειμένου να ευνοηθούν από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πιστεύουμε ειδικότερα για τους φόρους κατανάλωσης ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι η σωστή γιατί παρεμποδίζει μια καλύτερη κατανομή των εισοδημάτων. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ανεπίσημης και μη δεδηλωμένης εργασίας, είναι ένα ζήτημα ε, το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων ε, και συμφωνούμε με το ρόλο που μπορούν ε, να έχουν οι επιθεωρητές εργασίας του δουλευθέντος όμως γνωρίζουμε ότι με τις πολιτικές λιτότητας ε, είναι λιγότεροι και όχι περισσότεροι επιθεωρητές εργασίας και βλέπουμε λοιπόν ποια θα μπορούσε να είναι η σχέση μεταξύ των πολιτικών λιτότητας και των προτάσεων που ε, υποβάλλονται στο πλαίσιο του πακέτου αυτού. Όσον αφορά το θέμα των μισθών, ε, των αποζημιώσεων που για μας είναι μια, ένα κεφαλαιόδου σημασία ζήτημα και δύσκολο. Κάτι που πρέπει να μας ικανοποιεί στο πακέτο αυτό είναι ότι αναφέρεται στην πραγματική αύξηση των μισθών και απορρίπτεται στο εμέσως ε, ε, το πακέτο, ε, το, το κομμάτι που αφορά τις, τους ε, τους ε, μισθούς ε, στο πλαίσιο του πακέτου της απασχόλησης, όμως εξακολουθεί να αφορά ε, τους μισθούς ως ε, στοιχείο ε, ανταγωνιστικότητας θετικό και υποστηρίζει έτσι το γεγονός ότι για να είναι κάποιος ανταγωνιστικός πρέπει να μειώνει τους μισθούς. Κατά την άποψή μας αυτή, αυτό το μισθολογικό dumping είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για, για τα μέλη ε, της συνομοσπονδία μας ε, ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα το θέμα του βασικού μισθού. Για μας είναι ένα θέμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαπραγμάτευση των μισθών ε, στις ε, διάφορες χώρες. Για μας τίποτε δεν ε, αντικαθιστά τη διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των μισθών. Όμως, όπου χρειάζεται αυτό, ο ορισμός του ελάχιστου μισθού είναι κάτι το σημαντικό για να μπορέσουμε να μειώσουμε το, τη φτώχεια. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να συγχέεται ο αξιοπρεπής μισθός με τον ελάχιστο μισθό. Γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ελάχιστοι μισθοί οι οποίοι δεν είναι αξιοπρεπείς. Δεν επιτρέπουν δηλαδή ε, στους άνδρες και τις γυναίκες να διάγουν αξιοπρεπή βίο, ε, να έχουν παιδιά, να έχουν ένα διαμέρισμα και να ε, κάνουν τη ζωή τους όπως θα έπρεπε να μπορούν να την κάνουν. Υπάρχει ένας ε, αριθμός τομέων που αναγνωρίζονται ως τομείς που θα μπορούσαν ε, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης ε, στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα μιλάμε για τις πράσινες οικονομίες. Στους τομείς δηλαδή του περιβάλλοντος όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα θέσεων απασχόλησης. Για να μπορέσουμε όμως να εξορίξουμε αυτά τα κοιτάσματα θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις. Να υπάρξει μια χρηματοδότηση, άνευ της χρηματοδότησης, άνευ αυτών των κονδυλίων, αυτές οι θέσεις δεν μπορούν να ανέλθουν στην επιφάνεια και στο φως της ημέρας, να δημιουργηθούν ούτως ή πίν. Επομένως, ο στόχος αυτού του εγγράφου θα παραμείνει κάτι το οποίο θα είναι νεκρό γράμμα. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν τη σημασία του να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας στον κοινωνικό τομέα, στον υγειονομικό τομέα κτλ. ναι, πράγματι υπάρχουν δυνατότητες στον τομέα αυτό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις εδώ πέρα. Καταρχήν, αυτό είναι κάτι το οποίο εμπίπτει στον τομέα των κοινοφελών υπηρεσιών, των δημοσίων υπηρεσιών. Είναι δικαίωμα του καθενός να μπορεί να έχει υγειονομική περίθαλψη, να έχει πρόσβαση κοινωνικέ κοινωνικές υπηρεσίες και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το στόχο αυτό των κοινωνικών υπηρεσιών, των υγειονομικών υπηρεσιών, γενικά των δημοσίων υπηρεσιών να τις, να τις υπερασπιστούμε, διότι αυτή τη στιγμή προπυλακίζονται από τις τωρινές πολιτικές σε επίπεδο προϋπολογισμού στα κράτη-μέλη μας. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές, είναι οι τεχνολογίες της πληροφόρησης. Κάθε φορά εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι πιστεύω ότι δεν θα πρέπει <clears throat> να οδηγηθούμε μέσω αυτού του τομέα ο οποίος δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε μια νέα μορφή διαχωρισμού μεταξύ των ε, θέσεων εργασίας για τους άνδρες και των θέσεων εργασίας για τις γυναίκες. Οι γυναίκες κακοπληρωμένες δουλειές στον τομέα της φροντίδας και των υγειονομικών και της κοινωνικής περίθαψης και οι άνδρες στους τομείς που είναι καινοτόμοι και υψηλής τεχνολογίας. Αν θέλουμε να επιτύχουμε την αύξηση της απασχόλησης, αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να <clears throat> μην αυξηθεί το χάσμα αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών και να είναι οι γυναίκε μόνο στις κακοπληρωμένες δουλειέ. Για την κινητοποίηση των κοινοτικών ταμείων για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. προφανώς υποστηρίζουμε την κινητοποίηση αυτή των ταμείων, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αλλά πιστεύουμε ότι τα ταμεία αυτά θα πρέπει να κινητοποιηθούν και θα πρέπει να οδηγήσουν σε έργα τα οποία θα οικοδομηθούν μαζί με τους κοινωνικούς εταίρες, εταίρους για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών και στις ε, ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και κάθε περιφέρειας. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε να γίνονται πολλές πρωτοβουλίες αυτού του είδους. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν φυσικά όλα αυτά, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε, ιδίως σε χώρες όπως η Ισπανία που έχει τεράστιες δυσκολίες, όπως και η Ελλάδα, ότι αντί να προωθούνται οι πρωτοβουλίες αυτές, να χρησιμοποιήσουμε τον κοινωνικό διάλογο και τις κοινωνικές σχέσεις ως ε, τον κύριο άξονα αυτών των σχεδίων, τα σχέδια αυτά εκτιλήσονται έξω από τον κοινωνικό ιστό και τον κοινωνικό χώρο. Και αυτό με οδηγεί στο να σας είπω ότι η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου που προωθείται από το κείμενο αυτό <clears throat> είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε εντοπίσει κάτι το θετικό αλλά εξακολουθεί σε πολλές χώρες να βλέπουμε στην πράξη ότι συνεχίζεται μια επίθεση κατά των κοινωνικών σχέσεων και του, κατά του κοινωνικού διαλόγου. Όταν βλέπουμε ότι οι χώρες οι οποίες έχουν αντέξει καλύτερα στην ε, οικονομική κρίση είναι οι χώρες όπου είναι πιο εξελιγμένος αυτός ο κοινωνικός διάλογος. Και όταν βλέπουμε ότι από την άλλη πλευρά ότι οι πολιτικές της Τρόικας επιτίθενται εναντίον αυτού του κοινωνικού διαλόγου, το βλέπουμε αυτό στην Ισπανία, το βλέπουμε στην Ελλάδα, πρέπει τότε να κατανοήσουμε ότι υπάρχει <clears throat> μία κατά κάποιο τρόπο ε, διχοτομική μορφή διαχωρισμού μεταξύ λόγων και πράξεων, τουλάχιστον πράξεων σε αυτές τις χώρες που προανέφερα. Η πρόταση Κομισιόν επίσης μας φυστά την προσοχή μας για τα θέματα ευκυβερνησίας και οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Γίνεται μια πρόταση προς τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους για μεγαλύτερη συνεργασία. Ή αν θέλετε ε, μιας πιο έντονης διαβούλευσης γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό το θέμα του να υπάρχει μεγαλύτερη διαβούλευση. Εμείς όμως θεωρούμε ότι δεν είναι φυσιολογικό οι Υπουργοί Οικονομικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεδριάζουν, να συζητούν για τις αποδοχές των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανισότητες οι οποίες υπάρχουν, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ε, άνοδο της ένδυας, δεν θεωρούμε φυσιολογικό να οικειοποιούνται κατά κάποιο τρόπο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητήσεις για τις αποδοχές των εργαζομένων, χωρίς η σύνολη προβληματική της απασχόλησης να λαμβάνει υπόψη από αυτούς. Η προσπάθεια κατά συνέπεια του να συνδέσουμε τα θέματα της απασχόλησης με την συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση μας φαίνεται μεν θετική, αλλά πάντα επιμένουμε και θα επιμένουμε ότι το θέμα των αποδοχών δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο εθνικό από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και επομένως είναι κάτι το οποίο αρίεται της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συζήτηση για να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι μόνο σε σχέση με τις αποδοχές, αλλά και σε σχέση με τις ανισομέρειες <clears throat> προσφοράς και σύντησης. Η Συνομοσπονδία ε, εργατικών συνδικάτων στην Ευρώπη είναι έτοιμη να συζητήσει για τα θέματα αυτά, για τους μισθούς και τις αποδοχές. Τονίζουμε και πάλι ότι όλα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται από τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο εθνικό. Ίσως κάποια μέρα <clears throat> θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τους εργοδότες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι αύριο αυτή η μέρα. Να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι ότι σε επίπεδο διαβούλευσης έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα, διάλογο μακροοικονομικό ο οποίος μας προσφέρει ικανοποίηση σε πολλά επίπεδα. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει καταρχήν και επιπλέον ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω και να συμπεριλάβει όχι μόνο τους υπουργού Οικονομικών, αλλά και τους υπουργού Απασχόλησης, ώστε να μπορέσει να γίνει η σωστή σύνδεση μεταξύ απασχόλησης και οικονομικών και χρηματοοικονομικών. Τουλάχιστον αυτή είναι μια πρόταση που εμείς θα θέλαμε να διατυπώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> απαντώντας στο έγγραφο αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα ε, συγκληθεί το η εκτελεστικό μας συμβούλιο, θα παρουσιάσει τις προτάσεις Κομισιόν ο Επίτροπος Αντόρ και μετά από την εκτελε... τη συνεδρία Εκτελεστικής Επιτροπής Εκτελεστικού Συμβουλίου θα προκύψουν οι προτάσεις μας οι οποίες θα έχουν ένα χαρακτήρα δημόσιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αλεχάνδρο Σέρκας. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Σεγόλ για την πρώτη σας παρέμβαση και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα, είμαι μέλος των ε, σοσιαλιστών και θα ήθελα να αναγνωρίσω το ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων που καθημερινά δοκιμαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και ότι εσείς ε, δείχνετε μεγαλύτερη υπευθυνότητα αλλά και μεγαλύτερες απαιτήσει ε, ώστε να τηρηθούν οι αξίες και οι αρχές που βρίσκονται στην βάση στα θεμέλια της Ένωσης. Ε, είπατε και εμεί συμφωνούμε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία αλλά και ανησυχητικά προβληματικά στοιχεία στην ανακοίνωση και στα έγγραφα που την συνοδεύουν το πακέτο της απασχόλησης αύριο. Εμεί εδώ θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα όπου θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Αναγνωρίζουμε ότι το σύνολο των επιτρόπων έχουν μια νέα οπτική για τις δυνατότητες της Ευρώπης αλλά και για τις ανεπάρκειες αυτής και θα ήθελα να τον τονίσω ε, κάτι στη θέση μιας ε, βουλευτού που δεν είναι εδώ, της Ξηγιούτα Στέινρουκ, που είναι, ανησυχεί πάρα πολύ ε, για το θέμα των μισθών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο έγγραφο της Κομισιόν, που εισάγει ένα στοιχείο για τριμερή παρακολούθηση των μισθών, ενώ διαγράφει ένα μεγάλο κομμάτι της αυτονομίας και της βούλησης των ε, κοινωνικών εταίρων. Και μάλιστα με κάποιο τρόπο πιο υπόγειο, άλλες φορές όμως ε, και πιο βίαιο, να ενσωματώσει τη βούληση των κυβερνήσεων και των κράτων ε, για τα θέματα καθορισμού των μισθών. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ ανησυχητικό και ιδιαίτερα τη στιγμή που στην Ελλάδα βλέπουμε να καταπατώνται συλλογικές ε, συμβάσεις και εργατικά δικαιώματα. Να πω και δύο λόγια για το θέμα της νεότητας. Λίγο παραπάνω χρειάζεται από 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν ε, τόσα εκατομμύρια νέοι οι οποίοι δεν ε, φοιτούν κάπου και είναι άνεργοι. Πραγματικά ε, Πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα για να εγγυηθούν ε, το μέλλον των νέων. Πού θα βρουν τα χρήματα. Μάλιστα πολλά προγράμματα τελειώνουν και κλείνουν, ειδικά αυτά τα οποία βοηθούν τους πιο φτωχούς. Κάτι παραπάνω λοιπόν από ρητορικές εκφράσεις θέλουμε από πλευρά της Κομισιόν. Να τα δούμε δηλαδή όλα αυτά και με νομοθετικές προτάσεις και κυρίως με προτάσεις για τον προϋπολογισμό, για αύξηση των κονδυλίων. Να τελειώσω λέγοντας Δύο λόγια για την αναδιάρθρωση. Αύριο θα δουλέψουμε σε ένα intergroup για αυτό το θέμα. Για να περάσουμε δηλαδή από τα λόγια και πάλι στις πράξεις. Και τελευταία μου άποψη μιλάμε πολύ για το ρόλο των συνδικάτων. Εμένα με ανησυχεί πολύ μια αναθεώρηση που γίνεται στην μάλλον μια, ένας διαχωρισμός που γίνεται ανάμεσα στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης. Και αυτό γίνεται και μέσα στις πολιτικές οικογένειες. Γίνεται και στα συνδικάτα, συμβαίνει και στα συνδικάτα να ενσωματώνεται δηλαδή αυτός ο ιός της έλλειψης αλληλεγγύης Δηλαδή να σκέφτεται ο καθένα ότι όχι, οι άλλοι την έχουν πατήσει, αλλά εμεί δεν είμαστε σαν αυτού γιατί εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και το βλέπω τον ιό αυτό να έχει μολύνει διάφορες πολιτικές οικογένειες και ομάδες. Γιατί είδαμε τους Ιρλανδούς, είδαμε τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς και όλοι νομίζουν πως θα σωθούν. Ε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Alors, euh, Elisabeth Morin-Chartier et puis ensuite Ole Σαρτιέ και μετά. Ευχαριστώ πολύ κυρία τη Γενική Γραμματέα που ήρθατε σήμερα. Ε, στην Επιτροπή μας και να μας πείτε την άποψη των ε, Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για το θέμα αυτό του πακέτου απασχόλησης. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στο διάλογο αυτό να ε, αγγλίσουμε τις ιδέες μας αλλά και την ενέργεια που μπορούμε να ξοδέψουμε για την υπεράσπιση των θεμάτων αυτών, ειδικότερα λόγω της παγκόσμιας κρίσης, ε, η οποία πλήττει και την Ευρώπη με καταστροφικές συνέπειες για την απασχόληση. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ από την πλευρά της οικονομική, την οικονομική, τη χρηματοοικονομική και όχι τόσο πολύ από την κοινωνική πτυχή και κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνουν κοινωνικές ανακατατάξεις πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό το λόγο αυτό το πακέτο της απασχόλησης ε, πρέπει να το προσέξουμε, αλλά πρέπει στην Επιτροπή μας να μπορέσουμε να ε, ζητήσουμε και από τις υπόλοιπες ομάδες, από ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις υπόλοιπες επιτροπές, από ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας υποστηρίξουν σε αυτές τις ανησυχίες μας. Είναι ένα γενικότερο πολιτικό θέμα. Κάτι ακόμη, στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω, είναι το θέμα της πρόβλεψης. Εντάξει, δημιουργία των θέσεων απασχόλησης ε, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσληψιμότητα, αλλά ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις νέες θέσεις απασχόλησης και μάλιστα ένα επαγγελματικό κλάδο είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι μελέτες του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και διαφωτιστικές επί του θέματος αυτού. Βλέπουμε ότι αν προσθέσουμε ε, την ανάκαμψη της απασχόλησης με την ανανέωση των θέσεων απασχόλησης που έχουν να κάνουν με την κατηγορία της ηλικία ε, ε, και που συνταξιδοτηθούν, υπάρχουν πάρα πολλοί μισθωτοί ε, που μπορούμε να τους προετοιμάσουμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ε, ε, τα συνδικάτα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων να βοηθήσει με την εμπειρογνωμοσύνη της για την κάλυψη αυτού του κενού, κάτι που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το απαραίτητο για να μπορούμε να κάνουμε κάτι στην πράξη. Πώς λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αυτό που συζητούσαμε σε μια άλλη επιτροπή σήμερα για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Μπορεί να είναι ένα σημαντικό τομέα, εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις πράσινες θέσεις απασχόλησης πρέπει να βγούμε από τον τομέα του περιβάλλοντος ε, με τη στενή έννοια και να περάσουμε στον τομέα του κοινωνικού περιβάλλοντος, για να το πω έτσι. Ε, ποια είναι η δική σας εμπειρογνωμοσύνη από αυτού. Και το δεύτερο σημείο είναι τι είδους διακυβέρνηση για τα ευρωπαϊκά ε, κονδύλια ε, που ε, θα δαπανίσουμε για την ανάκαμψη της απασχόλησης σήμερα δεν χρησιμοποιούνται παρκώς, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια διαθέσιμα γιατί σήμερα αγωνιζόμαστε, η πρόεδρος το γνωρίζει πολύ καλά, για να υπερασπιστούμε ε, όλα αυτά τα κονδύλια και τη διάθεσή τους για την απασχόληση, αλλά εσείς ε, με το δίκτυο των κοινωνικών εταίρων σας πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να αναπτύξουμε προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των κονδυλίων αυτών, αλλά επιτρέπουν να είμαστε και πιο ε, αποτελεσματικοί. Υπάρχει λοιπόν και το πρόβλημα της διακυβέρνησης. Ένα τρίτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι η δημιουργία απασχόλησης. Βλέπουμε πολύ καλά βλέπουμε ότι δεν μπορούμε απλώς να υπερασπιζόμαστε θέσεις απασχόλησης για να προστατεύσουμε κάποιες θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να συνοδεύσουμε τις επιχειρήσεις ε, στην εξέλιξη, στην εξέλιξή τους. Ε, κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να σημαίνει την εξαφάνιση κάποιων θέσεων απασχόλησης και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι ε, με την ε, αξιοποίηση, με την ε, πιστοποίηση της, ε, των ικανοτήτων των δεξιοτήτων, να μπορέσουμε ε, τους ανθρώπους αυτούς εργαζομένους να τους προσαρμόσουμε σε ανάγκες επιχείρησης. Και γι' αυτό πρέπει να υποστηριχθούμε από τους κοινωνικούς εταίρους για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτήν την εξέλιξη και να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση εξαφάνισης της, ε, της θέσης εργασίας τους. Αναφερθήκατε επίσης ε, στις τεχνολογίες πληροφορικής ε, και επικοινωνίας και αντίθεση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εντάξει όμως πρέπει να προσέξουμε ότι το χάσμα αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτόν τον τομέα και μπορεί να είναι ε, ένα χάσμα και μεταξύ αστικών ε, περιοχών ε, και υπαίθρου και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι στην αντίδρασή μας, γιατί πάλι θα δημιουργήσουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, αστική και της υπαίθρου και οι, ε, πληροφο... οι τεχνολογίες πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, αν θέλουμε να επιτύχουμε μια ε, διακόπτει ε, η Πρόεδρος λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλοι ομιλητές ε, στον κατάλογο των ομιλητών, μα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχω να σας πω. Ε, καλά θέλετε να τα πείτε, αλλά μας τα λέτε το συνόρα. Πιστεύω λοιπόν ότι η κοινωνική εταίρη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να προβλέψουμε και ένα ποσοστό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε τους κοινωνικούς εταίρους σε όλες αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά η κυρία Σρότερ, η κυρία Ράπτη, η κυρία Μάρτιν, Νταρντέν, Μπενιό και εγώ ε, που θα ε, θέσω δύο ερωτήματα πάρα πολύ γρήγορα. Ε, κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Βερναδέτη Σεγκόλ για την γνωμοδότησή της για αυτό το πακέτο απασχόλησης. Έχει τονίσει ιδιαίτερα το ρόλο του δημόσιου τομέα. Έχει λοιπόν θέση στον πυρήνα του πακέτου αυτό. Τώρα, μέσα στο θέμα αυτό της απασχόλησης θα πρέπει να παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Μας είπατε κυρία Γενική Γραμματεύ ότι είναι δραματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αν εμείς επικεντρώσουμε την προσοχή μας μονάχα στην πράσινη οικονομία, στις πράσινες θέσεις απασχόλησης, στην πράσινη ανάπτυξη, στην προσπάθεια μιας ε, ε, πράσινης ανάπτυξης, έχουμε τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Εγώ ήμουν στο Χόρσενς στη συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ και βλέπω ότι πραγματικά γίνονται πολλές περισσότερες επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα από ότι στις ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτό είναι τελείως παράλογο αν θέλουμε να προετοιμάσουμε ένα πράσινο μέλλον. Για την ευελίξη ασφάλεια. Όπως είπατε, πολλές χώρες του Νότου θεωρούν ότι αυτή η έννοια είναι ουσιαστικά το να σε προσλαμβάνουν και μετά να σε πετάνε στον δρόμο. Όχι, η Δανία δεν έχει ένα τέτοιο σύστημα στην Δανία η ασφάλεια είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε. Δεν είναι η κυβέρνηση που καθορίζει τι περιεχόμενο θα έχει η ασφάλεια. Γι' αυτό λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα μα. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι θετικό. Το να μπορούν να συζητούν οι κοινωνικοί εταίροι και επίσης να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια και να συζητούν για το μέλλον της εργασιακής αγοράς. Πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα μεν, αλλά δεν μπορεί να είναι μονάχα κάτι του οποίου την ύφη θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία στην εργασιακή αγορά, αλλά για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε τι μορφές απασχόλησης, όπως είναι μερική απασχόληση ή οτιδήποτε τέτοιο, θα πρέπει να <clears throat> χρησιμοποιηθούν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Νότια Ευρώπη που δεν έχουν ποτέ ένα σταθερό συμβόλαιο. Θα πρέπει η ευελιξία αυτή να συνοδεύεται από κάποια βεβαιότητα, από κάποια ασφάλεια. Και όχι να είναι μονάχα επιβολή περισσότερων φόρων. Είναι απαραίτητο να έχει κανείς αποδοχές οι οποίες του επιτρέπουν να επιβιώσει, να πληρώνει τους λογαριασμούς του στο τέλος του μήνα. Αλλιώς γιατί να πηγαίνει να δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική απασχόληση η οποία να είναι ενεργή και επίσης μια πολιτική ε, κατάρτισης και παρακατάρτισης για να μπορεί να αλλάξει κανείς μορφή εργασίας. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλα στοιχεία στο πακέτο αυτό ή καλύπτει αρκετά όλα αυτά τα ζητήματα που θέλουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σεγκόλ για την εισήγησή της. Πραγματικά ευχαριστώ, μαζί, ε, συμφωνώ μαζί σας ε, όσον αφορά τα διάφορα μέτρα λιτότητας που έχουν φέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι η ανεργία στην Ελλάδα και μετανάστευση των ανθρώπων ε, σε ηλικία εργάσιμη έχει αυξηθεί. Επίσης η μαύρη οικονομία αναπτυχθήκε και αυτά είναι τα αποτελέσματα λιτότητας ανεφλόγου. Τώρα πρέπει λοιπόν να ξανακοιτάξουμε την ανάπτυξη, την προώθηση της της οικονομίας και την απασχόληση. Συμφωνώ πως σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για ορισμένες πτυχές της πολιτικής απασχόλησης του. ωστόσο θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα της ε, ευελεξασφάλειας. Πιστεύω πως ο ανταγωνισμός προωθείται όταν έχουμε ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια. Ωστόσο, ε, συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες. Για παράδειγμα, στη χώρα μου η κυβέρνηση πρότεινε ένα πακέτο κανόνων για την απελευθέρωση των εργατικών ε, ε, σχέσεων, διότι μόνο λέει, η απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά μας. Για παράδειγμα, χαμηλότερη ασφάλεια για τους συνταξιούχους, για τους νέους, για τους ανάπηρους, για τις γυναίκες, Οπότε Πιστεύω πω τα, τα συνδικάτα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρά στην αξιολόγηση του τέτοιων μέτρων. Η ευελιξασφάλεια μπορεί να, να λειτουργήσει στη Δανία και στι κάτω χώρε, αλλά πρέπει να προσέξουμε πολύ σε άλλα κράτη-μέλη όπω η Ιρλανδία όπου η κοινωνική εταίρεια είναι τόσο ισχυρή. Για παράδειγμα, έχουμε 70, στην Δανία 70% μόνο στα συνδικάτα, ενώ εμεί έχουμε 10% των εργαζομένων στη Λιθουανία που ανήκουν σε συνδικάτα ο λαός μας λοιπόν υποφέρει από αυτή την ευέλικτη ασφάλεια. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω και για το θέμα των ελάχιστων ημερομηνιστήρων. Σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει αυτό το, το ανεπίλητο πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια και πολλοί κόσμος που λαμβάνει το μήνυμο ε, μισθό τώρα είναι κάτω από το επίπεδο της στόχιας και είναι ε, παγιδευμένοι σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με εμπειρογνώμονε και να βρούμε ποιε είναι οι προτάσεις από, από εδώ, από το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να πληρούνται κάποια κοινά κριτήρια για του ελάχιστους ελάχιστους μισθούς. Ähm, Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Σουέντερ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ένα σημαντικό θέμα είναι το θέμα των πρασίνων θέσεων απασχόλησης. Από την άποψή μας γίνεται σαφές από το κείμενο ότι το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τη σημασία αυτών των θέσεων εργασία. Όχι μόνο να έχουμε λοιπόν μία χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά να έχουμε και το κατάλληλο πλαίσιο. Βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία ότι λόγω των νέων συνδικών εργασία στην ε, Γερμανία πολλέ θέσει εργασία έχουν καταστραφεί γιατί δεν υπήρχαν οι απαραίτητε προποθέσει, το απαραίτητο πλαίσιο. Έχουμε νέε επιχειρήσει οι οποίες έχουν πολύ καλές ιδέες, έχουν ευρεσιτεχνίες, αλλά τελικά δεν τα βγάζουν πέρα γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουν τα, το απαραίτητο πλαίσιο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε όχι μονάχα να υπάρχουν τα νέα στοιχεία, αλλά να μπορέσουν να διατηρηθούν και οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας που υπάρχουν παραγωγή χάρη στην οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης θα ήθελα να γνωρίσω ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα, τη... η... θα αναλάβουν τα συνδικάτα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τίθεται το θέμα των ελαχίστων μισθών. Και νομίζω ότι οι πρωτοβουλίε οι οποίε βρίσκονται σε αυτό το πακέτο δίνουν την ευκαιρία στα ευρωπαϊκά συνδικάτα να ξεκινήσουν μια εκστρατεία στην Ευρώπη ώστε να υπάρξει ένα επαρκές επίπεδο ελαχίστων αποδοχών για όλη την Ευρώπη ο οποίος να βρίσκεται στο επίπεδο του μέσου εισοδήματος. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχέδια για μια τέτοια καμπάνια στην εκτελεστική σας επιτροπή. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αν μπορείτε να σκεφτείτε με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για να υπάρξει και προβληματισμός για το θέμα αυτό, όπως πρέπει να υπάρξει και στο δικό μας κοινοβούλιο. Και το τονίζω αυτό γιατί πράγματι εγώ νιώθω αποτροπιασμό για το γεγονός ότι υπήρξε παρέμβαση στην Ελλάδα στα θέματα των κατοτάτων αποδοχών και εγώ το θεώρησα αυτό μια άμεση προσβολή των δικαιωμάτων των συνδικάτων στην Ευρώπη και πιστεύω ότι δεν έχει υπάρξει αρκετή προβληματική στην Ευρώπη για αυτή την επίθεση κατά των εργαζομένων. Η κυρία Ράπτη, η οποία νομίζω μπορεί να συνεχίσει στο θέμα αυτό με την Τρόικα και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Σεγκόλ. Είναι χαρά να την έχουμε κάθε φορά εδώ. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλήτρια. Ε, αυτή τη φορά θα διαφωνήσω λίγο μαζί της. Ε, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία της για το έγγραφο της Κομισιόν. Και αυτό γιατί έχουμε δει μέχρι τώρα ότι έγγραφα της Κομισιόν, τα οποία περιλαμβάνουν α, ποινές και επιβολές όρων πάντοτε εφαρμόζονται. Έγγραφα της Κομισιόν, τα οποία βλέπουν με θετικότερο μάτι την απασχόληση, πάντοτε μένουν έγγραφα. Δεν γίνονται ποτέ πράξη. Άρα φοβάμαι. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την αξιοπρεπή εργασία. Ο όρος «decent work» ήταν α, μέσα σε κάθε πρόταση που συζητούσαμε σε αυτή την Επιτροπή. Στα τρία σχεδόν χρόνια που βρίσκομαι εδώ, ο όρος «decent work» σταματάει πια να εμφανίζεται, κοντεύει να εξαφανιστεί. Και βεβαίως καταλαβαίνω ότι αυτό έχει σχέση με αυτό που αναφέρατε, το «decent wage». Ε, το ερώτημά μου είναι για σας, για τα συνδικάτα ποιο είναι το περιεχόμενο του decent work. Υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει ή πρέπει να το ξαναδούμε και σε ποια όρια θα τοποθετηθεί. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι εάν η, η θέση που έχετε απέναντι στο έγγραφο της Κομισιόν ε, είναι ομόφωνη από, την Ένωση των Συνδικάτων ή όχι. Και αυτό για μένα έχει σημασία γιατί όπως προανέφερε ο συνάδελφος Σέρκας αρχίζουμε να έχουμε διαχωρισμούς βορρά-νότου και μέσα στα συνδικάτα. Και θεωρώ ότι είναι τεράστια σημασίας το γεγονός ότι τα συνδικάτα πρέπει να μένουν ενοποιημένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η άμυνα των εργαζομένων όλης της Ευρώπης. Ε, τέλος, πράσινες θέσεις εργασίας. Πριν δημιουργηθούν οι πράσινες θέσεις εργασίας, θέλω να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας. Γιατί στις παραδοσιακές θέσεις εργασίας παρατηρούνται συνεχώς απολύσεις. Στις δε πράσινες θέσεις εργασίας πολύ σωστά επισημάνατε, χρειάζονται επενδύσεις. Για τις επενδύσεις χρειάζονται χρήματα και χρήματα δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι συζητάμε με πολύ καλή διάθεση πάνω σε ένα έδαφος που τρέμει όπως τρέμει και το έδαφος της Ιταλίας τον τελευταίο καιρό από τους σεισμούς. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Χάρκιν και ο κύριος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους και στην κυρία Σεγκόλα. Έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια. Καταρχήν είπατε ότι αυτό το πακέτο δεν μπορεί να λειτουργήσει αν είναι παράλληλα με την λιτότητα, αν συνοδεύεται από λιτότητα. Εμείς στην Ιρλανδία προσπαθούμε κάπως να τα διαχειριστούμε και τα δύο αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ θα φτάσει στα 120% ε, που είναι αβάσταχτο και ταυτόχρονα προσπαθούμε κάπως να σταθούμε εξελιχθούμε ως χώρα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό να μπορούμε να ξαναπάμε και να ξαναδανεστούμε από τις αγορές, αλλά ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούμε και επασχόληση. Πιστεύω λοιπόν ότι σε εθνικό επίπεδο ε, κλαίγουμε τις ε, κυβερνήσεις μας για ώστε αυτές να προβαίνουν σε επιλογές για το πώς δαπανούν τα χρήματα και ενώ μπορείς να έχεις κάποιο επίπεδο λιτότητας, εξαρτάται ποιον θα χτυπήσει αυτό και πώς ε, και αν βλέπεις ε, τη φορολογία ως μέθοδο συλλογής εισοδημάτων ή ε, αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα επίπεδα και μπορώ να πω ότι μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Όταν είναι άκαμπτη η κατάσταση και δεν υπάρχει ευελιξία, ναι, δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί μέσα σε όλα αυτά. Και θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Μιλήσατε επίση για τα διαρθρωτικά μέσα και είπατε ότι στην ουσία ασχολούμαστε με την, ε, ε, ζήτηση, με την προσφορά και όχι με τη ζήτηση. Πώς μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε και να κινητοποιήσουμε την πλευρά της ε, ζήτησης. Τώρα, για την ευελιξασφάλεια είπατε ότι κάποιες χώρες είναι καλύτερες και άλλες όχι τόσο καλές και είπατε για το κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα και την Ισπανία και είναι πολύ κρίσιμο αυτό. αλλά υπάρχουν άλλα παραδείγματα κατά τη γνώμη σα σε άλλες χώρες όπου το θέμα τη ευελιξασφάλεια δεν πάει καλά πέρα από τον κοινωνικό διάλογο βέβαια που θεωρώ ότι είναι όντως σημαντικός. Και έχω μια διαφορά όσον αφορά την ε, κοινή βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ε, Βέβαια, ο λόγος είναι ότι πολλές από, πολλοί από αυτού τους φόρους θα πάνε στις μεγαλύτερες οικονομίες, ακόμα από μια μικρή εξαγωγική χώρα, γιατί αυτοί είναι που θα καταναλώνουν τη ε, αγαθά αυτά. Πολλοί εργαζόμενοι λοιπόν στην Ιρλανδία θα διαφωνούσαν μαζί σας για το συγκεκριμένο σημείο, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση. Και κάτι ακόμα. Είπατε ότι ότι οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν καταλάβει όλε τι συζητήσει, ε, μονοπολούν τι συζητήσει, Έχετε δίκιο και εγώ υποστήριξα τις τη Λισαβόνα, χάρη στο άρθρο 9. Εδώ όμως ε, σε αυτή την περίσταση η κοινωνική ρήτρα απλώ δεν εφαρμόζεται. Ε, θα μπορούσε και να μην υπάρχει καθόλου. Χάνουμε λοιπόν αυτή την ισορροπία και εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και να εξασφαλίσουμε την επιστροφή αυτή τη ισορροπία. Και τέλο έχει λάβει κάποια θέση η TUC όσον αφορά την συνθήκη και πώς θα πρέπει να ψηφίσουν ε, οι Ιρλανδοί επ' αυτής. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Γενική Γραμματέα για την παρουσίασή της και τα διάφορα σχόλια αυτά. Νομίζω ότι το πακέτο για την απασχόληση είναι μια ευκαιρία και ναι. χαίρομαι που η Κομισιόν έχει παρουσιάσει μια τέτοια πρόταση. Εγώ ναι. είμαι πολύ κοντά στις προτάσεις σας και αυτό φαίνεται και από τους τροπολογίες μου στις διάφορες εκθέσεις που εγώ παρακολούθησα. Θέλω να κάνω λοιπόν ορισμένα σχόλια. Πρωτού φτάσω <clears throat> στα ερωτήματά σας. Είπατε ότι η βία λιτότητα δεν βοηθάει <clears throat> στην ε, επίτευξη θέσεων απασχόλησης, ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με προβλήματα όπως η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Δεν πρέπει επίσης, όπως σωστά υπογραμμίσατε, το θέμα αυτό να αφαιθεί μονάχα στους Υπουργούς Οικονομικών. Πρέπει να εμπλακούν και οι Υπουργοί Απασχόλησης, οι Υπουργοί Κοινωνικών Υποθέσεων. Αλλά με λιγάκι ή ίσως δεν κατάλαβα καλά τη θέση σας σε σχέση με τους κατώτατους μισθούς. Βλέπουμε να φοβάστε κάπως να είσαστε διστακτικοί σε σχέση με αυτή την πρόταση που για μένα θα ήταν θετική όταν μιλάει η Κομισιόν για κατώτατους μισθούς. Όταν λέτε ότι δεν πρέπει να αντικαταστήσει τους μισθούς που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ότι δεν πρέπει να την συγχαίουμε με μια αξιοπρεπή, με αξιοπρεπούς, αξιοπρεπείς μισθούς, ότι πρέπει να είναι ένα εθνικό θέμα μέσα στα πλαίσια της έκθεσης για τον αγώνα κατά της ένδυας. Θυμάμαι ότι είχατε αγωνιστεί υπέρ του ελάχιστου εισοδήματος. Προφανώς αυτό είναι διαφορετικό, αλλά το ένα μπορεί να φέρει το άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να υπάρξει η έννοια του κατώτατου μισθού και είναι μια πρόοδος αυτό. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν γιατί έχετε μια τόσο διστακτική θέση. Ποιοι είναι οι φόβοι σας. Και τώρα το θέμα της ΆΤΑ, της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Ξέρετε ότι αυτό στο Βέλγιο είναι ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα και χαίρομαι που στο πακέτο για την απασχόληση και στην ε, παρέμβασή σας ότι πρέπει να προωθήσουμε την αρχή της πραγματικής αύξησης των ε, αποδοχών, ε, δηλαδή πέρα από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Τότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να προωθηθεί ένα τέτοιο σύστημα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Ο κύριος Μπενιό ο Πουπάκης και ο κύριο Φαλ, κλείνω τον κατάλογο των αγορητών, αλλά προηγούμενος ο κύριος Φενιό. Ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα με ενδιαφέρει και μιλάω για την ενίσχυση της ζήτησης στην οικονομία. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε, διέρεσης μεταξύ της ε, ανάπτυξης, της απασχόλησης από τη μία και από την άλλη ε, της λιτότητας. Ε, κάποιοι είναι επιφυλακτικοί, αλλά από την άλλη πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα λιτότητα, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα και δεν είναι δυνατόν να το παραγνωρίσουμε και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε και με αυτή την κατάσταση. Οπότε το πρόβλημα είναι να δημιουργηθεί ζήτηση στην οικονομία και αυτό δεν είναι κάτι απλό να γίνει. Πρέπει να ε, κάνουμε στοχευμένες προσπάθειες. Ε, μόνο δύο-τρία κράτη-μέλη έχουν ε, την επιλογή μιας δημοσιονομικής ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Δεν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα πολλών κρατών μελών. είναι αυτό που κάνει το, το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα. Ε, μπορεί να υπάρχει μια πληθωριστική τάση λόγω αυτού, αλλά ε, φαντάζομαι ότι υπάρχει τρόπος να το διορθώσουμε αυτό. Το μόνο πρόβλημα λοιπόν με αυτήν την τη δημοσιονομική ενίσχυση είναι κάπως ε, να προσπαθήσουμε να ε, στοχεύσουμε την ε, χρηματοδότησή μας σε τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση στην οικονομία, όπως είπα. Αν χρειάζεται λοιπόν να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα εκεί, από κάπου αλλού πρέπει να περικόψουμε. Όμως αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ανάπτυξης της ζήτησης, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, δεν ε, σημαίνει ότι σε δύο-τρία χρόνια θα δούμε τα πρώτα ε, αποτελέσματα. Ε, όλοι λένε ότι θέλουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά κανένας δεν μας λέει ποιο ακριβώς είναι το, το πρόγραμμα αυτό. Δεν μπορεί κανείς να συνεχίσει να δανείζεται όταν έχει ήδη δανειστεί πολύ. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες ε, ε, φορολογικού τύπου αλλαγές, ε, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα έσοδα αυτών που πληρώνονται περισσότερο, όχι να τους δίνουμε περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο ενίσχυσης της ζήτησης, μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας προσέγγισης. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν ακούστηκαν αρκετές ερωτήσεις, ε, κυρία Σεγκόλ, θα προσθέσω και εγώ δύο. Το πρώτο είναι... Ποια είναι η άποψή σας για τις συστάσεις αναχώρα που μόλις δημοσίευσε σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχατε τη δυνατότητα ίσω, όπω άλλωστε ούτε και εγώ να δείτε τις ε, λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να μας πείτε ορισμένα πράγματα όσον αφορά τον επαναπροσανατολισμό ε, των πολιτικών ε, υπέρ τη συζήτηση, όπως κάποιοι εξημών εδώ σα συζητούν. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι το θέμα του μακροοικονομικού διαλόγου, γιατί στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και του εξαμήνου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού αυτό. Ε, είπατε πολλές φορές ε, ε, και το έχουμε συζητήσει και με προκατόχους σας, είναι καθαρά επίσημο, έχετε πει ότι το έχουμε κάνει, οπότε όλα πάνε καλά, όμως δεν είναι ο πραγματικός μακροοικονομικός διάλογος που τον έχουμε ανάγκη. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποτέ δεν έχουμε προσκληθεί ούτε ως παρατηρητές. Μήπως έχετε καμιά ιδέα πιο συγκεκριμένη για το τι θα έπρεπε να ζητήσουμε γιατί μερικές φορές ε, ε έρχεστε να μας βοηθήσετε και εμείς ευχαρίστω ως εξωτερικοί παράγοντες να σας, να σας βοηθήσουμε σε αυτόν τον διάλογο τον μακροοικονομικό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ε, ζητήθηκε για παράδειγμα η Επιτροπή Οικονομικών και Απασχόλησης να συμμετέχουν ε, σε αυτή την προσπάθεια. Ένα τέταρτο έχετε για να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ θα σηκώσω το γάντι. Θα αντιμετωπίσω την πρόκληση αυτή, ξεκινώντας και βέβαια δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όλες τις ε, παρεμβάσεις. Θέλω να σταθώ στα σημεία που μου φαίνονται μείζωνα για τις διάφορες, παρεμβα... στις διάφορες παρεμβάσεις. Να σας πω καταρχήν ότι δεν έχουμε διαφορές απόψεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κρίση. Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την κοινότητα απόψεων που υπάρχει μεταξύ των χωρών που είναι σε καλύτερη θέση αν θέλετε μέσα στην ε, Ομοσπονδία Συνδικάτων, δηλαδή τη Γερμανία και τις χώρες της ισχυρής οικονομίας και αυτές οι οποίες είναι λιγότερο, <clears throat> σε λιγότερο καλή θέση λόγω των πολιτικών λιτότητος. Την ίδια θέση έχουμε. Λέμε όλοι από κοινού ότι αυτές οι πολιτικές μας έχουν φέρει σε ένα αδιέξοδο και μας έχουν ουσιαστικά κολλήσει στη γωνιά και δεν μπορούμε να βγούμε από εκεί αν δεν τις αλλάξουμε. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το έγγραφο αυτό που έχω ενώπιόν μου και εσείς δεν το έχετε ακόμα στα χέρια σας. Είναι ένα έγγραφο το οποίο ακόμα δεν έχει εγκριθεί από την εκτελεστική μας επιτροπή θα γίνει αυτό την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να σα το δημοσιοποιήσω λοιπόν το έγγραφο αυτό, παρά το γεγονό ότι νομίζω ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένο, ώστε αυτέ οι οδηγές γραμμέ του που σα παρουσίασα να είναι σίγουρο ότι θα υποστηριχθούν και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά το ίδιο το έγγραφο δεν θα δημοσιευτεί παρά μόνο την επόμενη εβδομάδα και αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τους κανόνες της συνδικαλιστικής δημοκρατίας που είναι σημαντικές στον φορέα μας. Ένα άλλο θέμα που μου ετέθη ευθέως πολλές φορές είναι το θέμα του κατώτατου μισθού. Όχι του κατώτατου εισοδήματος, αλλά του κατώτατου μισθού. Γιατί θεωρήσατε, <clears throat> μου είπατε, δισταγμούς σε αυτά που είπα. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν διαφορετικά συστήματα λειτουργίας των κατώτατων μισθών. Έχουμε μία σειρά χωρών όπου το θέμα του κατώτατου μισθού κινδυνεύει να παρακάμψει την ε, αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τη δυνατότητά τους να καθορίσουν τις αποδοχές του εργαζομένου. Αν λοιπόν <clears throat> αυτές οι χώρες μπορούν να προστατεύσουν τις αποδοχές των εργαζομένων με τις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Λέμε όμως επίσης στην Συνομοσπονδία Συνδικάτων ότι στις χώρες που είναι απαραίτητο και το ζητούν τα συνδικάτα να υπάρχει κατώτατος μισθός, αυτός ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να δημιουργηθεί ή να αυξηθεί. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα μία σαφής απόφαση, εμείς θέλουμε να κινηθούμε προς ένα κατώτατο μισθό, ο οποίος θα έχει το χαρακτήρα ενός ποσοστού, θα είναι πάνω από 50% των μέσων αποδοχών τίνοντας προς τα 60% ή τουλάχιστον 60% του μέσου μισθού. Αυτά είναι λοιπόν <clears throat> του μισθού μάλλον που 50% των εργαζομένων έχουν πάνω από αυτόν. Αυτό μας ευθυγραμμίζει με τις θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα επιτρέψει σε χώρες που έχουν πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό να αυξήσουν αυτό το κατώτατο μισθό Προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχουν λοιπόν καθόλου δισταγμοί σε σχέση με τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από την εισαγωγή ενός κατώτατου μισθού. Εκεί που το θέλουν τα συνδικάτα υπάρχει σίγουρα μια μορφή δισταγμού <clears throat> για τις χώρες που είναι διαφορετική διαδικασία καθορισμού των μισθών και όπου οι αποδοχές καθορίζονται αποκλειστικά από διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα <clears throat> να προσθέσω ότι για το θέμα αυτό πιστεύουμε ότι είναι σαφές για μας ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια μεγαλύτερη προετοιμασία, μια διαδικασία διαβούλευσης με τα συνδικάτα προτού καταλήξουμε σε ένα ελάχιστο μισθό. Έρχομαι τώρα σε όλα τα θέματα της ευελίξης ασφάλειας. Δεν θέλω τώρα να σταθώ υπερβολικά στο σημείο αυτό. Θέλω να επιμείνω έντονα στο ότι είναι σαφές για μας ότι στο βαθμό που υπάρχει ασφάλεια της απασχόλησης, ασφάλεια για τις περιόδους <clears throat> ε, ανεργίας, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε την έννοια της ευελιξίας. Υπάρχει αυτό στη Δανία. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει βέβαια και η Δανία ακόμα ορισμένα προβλήματα, αλλά σίγουρα ένα τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ευέλιξη ασφάλεια σε ένα εργαζόμενο που ξέρει ότι μπορεί την επόμενη εβδομάδα να τον πετάξουν από τη δουλειά του και μετά δεν θα έχει καθόλου εισόδημα, αυτό δεν είναι σοβαρό. Αυτό σημαίνει απλώς ότι του πουλάμε την ευελιξία και χωρίς καμιά ασφάλεια. Μπορεί λοιπόν για ορισμένε χώρε να είναι αυτό μια θετική αντιμετώπιση, μια θετική διαδικασία, αλλά αναπόφευκτα για πάρα πολλές άλλες χώρες η έννοια της ευέλικης εξαντλείται, διότι την κατανοεί κανείς μονάχα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια και να μιλάμε απλώς για μια ενεργή εργασιακή πολιτική με τη βοήθεια των κονδυλίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Για όλα τώρα τα θέματα, τα οποία άπτονται της ανάπτυξης και της λιτότητας. Να είμαστε σαφείς. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων λέει ότι θα πρέπει πράγματι να εξασφαλίσουμε, να επανέλθουμε σε μια επανεξισορρόπηση των δημοσίων οικονομικών και σε μια εξυγίανσή τους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την εξυγίανση αυτή. Το θέμα είναι πώς. Μπορούμε να μειώσουμε το χρέος των κρατών μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η απάντησή μας είναι όχι. Είναι πιθανό και πολύ πιθανό ακόμα για μας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανάπαυλα στις πολιτικές λιτότητες, οι οποίες τελικά αύξησαν το κρατικό χρέος. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Απλώς αυξήθηκε το χρέος των χωρών αυτών. Θα πρέπει να υπάρξει μια ανάπαυλα για να υπάρχει μια ευκαιρία για την ανάπτυξη. <clears throat> για μας είναι και θέμα λοιπόν χρόνου και χρονισμού. Κάτι ακόμα πρέπει να σας πω και το οποίο το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Είναι πολύ πιο δύσκολο να επαναφέρουμε την ισορροπία, την κοινωνική ισορροπία μιας χώρας από ότι να επαναφέρουμε την ισορροπία σε επίπεδο προϋπολογισμού. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε μια χώρα να ανατρέψει την κοινωνική ισορροπία και είναι πολύ δύσκολο να την επανέβρει. Και νομίζω ότι σε ορισμένες χώρες έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. για το ερώτημα που μου θέσατε. από, τον, από το μέλος του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ήταν εναντίον του Δημοσιονομικού Συμφώνου γιατί θεωρούσαμε, θεωρήσαμε ότι είναι και περιττό και δεν θα επιτύχει το στόχο του. Κατανοούμε όμως τις δυσκολίες των επιλογών για την Ιρλανδία. Γνωρίζουμε ποιες είναι θέσεις Ιρλανδικής Νομοσπονδίας Εργατικών Ενώσεων, της οποίας τα μέλη βρίσκονται μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Τους λένε ότι εάν δεν υπογράψετε αυτό το σύμφωνο δεν θα έχετε πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια, επομένως τι θα γίνει τότε στη χώρα σας. Και υπάρχουν οι άλλοι που λένε ότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να μας βοηθήσει σε τίποτα αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο. Δεν είναι ούτε η πρόθεσή μου, ούτε είναι δική μου αρμοδιότητα να επισέλθω στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα συνδικάτα σε εθνικό επίπεδο. Εγώ έχω απόλυτο σεβασμό για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ιρλανδοί συνάδελφοί μας για το θέμα αυτό και για τη θέση που έχουν, θα έχουν σε σχέση με το δημοψήφισμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα τόνωσης της ανάπτυξης. Έχουμε μιλήσει για τη χρήση των κοινωνικών ταμείων, <clears throat> για την ανάγκη να εκμεταλλευτούμε τον κοινωνικό διάλογο και εδώ θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο, αλλά μάλλον μένω από χρόνο, αλλά ας είμαστε σοβαροί. Είναι δυνατόν πέραν των ευρωμολόγων, πέραν μια εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του ευρώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε επαρκή εμπιστοσύνη στο ευρώ, ώστε να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν αυτές οι επενδύσεις και να επιτρέψουμε αυτήν την ανάπτυξη. Η απάντηση είναι όχι και συμφωνώ με αυτούς που, που Λένε ότι κάποια εκατομμύρια ευρώ για, αλλά για τον καθένα μας χώρια είναι πολλά τα εκατομμύρια αυτά αλλά πάντως δεν θα επηρεάσουμε την απασχόληση με κάτι ψώρο εκατομμύρια Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα λοιπόν, ένα όραμα αποφασιστικό για το πώς θα βγει η Ευρώπη από από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιάλθει. Αλεσάνδρο, ξέρετε πολύ καλά ότι τη Γιωσή εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι υπέρ ενός νομικού πλαισίου σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις και ότι πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τις αναθεωρήσεις, της νέες, ε, θέσεις απασχόλησης ε, και τα λοιπά, θα πρέπει φυσικά να αναπτύξουμε την μόνιμη παιδεία και κατάρτιση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με μια χρηματοδότηση και μια χρηματοδότηση που είναι σημαντική, σημαντική και δεν θα τη βρούμε, δεν την έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, για τις συγκεκριμένες ε, συστάσεις αναχώρα δυστυχώς δεν μπόρεσα. Δεν προτιμώ μάλλον να μην πω τίποτα για την ώρα, γιατί δεν είχα το χρόνο μέσα στην ημέρα σήμερα να το διαβάσω όλα αυτά με τους διάφορους συμβούλους, οικονομολόγους, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω απάντηση σύντομα. Όσον αφορά τον μακροοικονομικό διάλογο, συμφωνώ απολύτως για, για την ώρα είναι ε, κάτι το τυπικό. Βέβαια υπάρχει, κάτι είναι και αυτό. Εμείς αυτό που προτείνουμε για τον μακροοικονομικό διάλογο είναι περισσότερες ανταλλαγές ανάμεσα στους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, τους Υπουργούς Οικονομικών και Απασχόλησης, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό θα έπρεπε οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία που αφορά την ε, έλλειψη μακροοικονομικής ισορροπίας, τους ε, πίνακες, ε, τους μηχανισμούς η προειδοποίησεις και της αναχώρα ανάλυσης. Μόνο αν αυτός ο διάλογος και η προηγούμενη αυτή προπαρασκευή θα μπορέσει να οδηγήσει στο να είμαστε πιο παραγωγική και αποδοτική. Euh, Στα πόσα λεπτά είμαι πρόεδρε δεν ξέρω. Για δύο λεπτά να δω τις σημειώσεις μου. Για τις πράσινες θέσεις επασχόλησης, ε, η Ελίζα Σρέντερ με ερώτησε, χρειάζονται επενδύσεις μεγάλων διαστάσεων. Συχνά έχουμε οθήσει και αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να εμβαθύνουμε ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για παράδειγμα τη μεταφορά της ενέργειας ε, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες ε, από χώρες όπου η ενέργεια αυτή είναι πιο προσβάσιμη. Αλλά και πάλι αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, τα μεγάλα αυτά προγράμματα είναι διαθέσιμα μόνο σε μακροοικονομικές συνθήκες οι οποίες για την ώρα δυστυχώς δεν πληρούνται. Τέλος, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κοινωνικό διάλογο, όλοι συμφωνούν για τον κοινωνικό διάλογο. Είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιον που θεωρητικώς διαφωνεί με τον κοινωνικό διάλογο. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα στη Λιθουανία ξέρω πάρα πολύ καλά το τι γίνεται με τον κοινωνικό διάλογο και όχι μόνο στη Λιθουανία. Οι Ισπανοί συνάδελφοι μου λένε ότι διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία με τους εργοδότες που αμέσως μετά ε, καταργήθηκε μέσω μιας κυβερνητικής απόφασης αλλά ο, κοινωνικό ο κοινωνικός διάλογος ε, πάει για βρούβες, με συγχωρείτε και για την έκφραση. Ε, θα πρέπει λοιπόν ναι, να στηριχθεί ο κοινωνικός διάλογος και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γι' αυτό. Τώρα για την αυτόματη αναπροσαρμογή ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της αυτόματης αναπροσαρμογής, της αριθμικής αναπροσαρμογής στο Βέλγιο και πώς επιτρέπει στους πραγματικούς μισθούς να μένουν ε, στο, σε συγκεκριμένη θέση. Αλλά μην μου ζητάτε να ζητήσω και αυτό. Θα ήταν καλό να διευρυνθεί, αλλά για την ώρα θα ήταν πολύ δύσκολο για μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά οι Βέλγοι και όσοι έχουν ακόμα την ΆΤΑ έχουν όλοι μας τη στήριξη και να τη διατηρήσουν εκεί όπου βρίσκεται. Δεν ξέρω να απάντησα σε όλα τα ερωτήματα, πάντως προσπάθησα. Πάντως, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η τελευταία σας απάντηση, από ό,τι κατάλαβα. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι δεδομένου του αριθμού των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν, αλλά νομίζω πως υπήρξε έτσι μια πλούσια ανταλλαγή απόψεων που απηχεί και άλλες εργασίες που κάνουμε εμείς εδώ. Νομίζω ότι πολλά μηνύματα πέρασαν και ότι θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια με τους συνεργάτες ε, σε διάφορα θέματα να επανέλθουμε. Ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συμμετοχή σας ε, και στο επανειδήν. Euh, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν έρθει ο επίτροπο Ζαντορ, σα προτείνω να αρχίσουμε τη συζήτηση για το σημείο 11 και όταν ε, καταφτάσει ο επίτροπο, να σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Για το σχέδιο της προφορικής ερώτησης και το κείμενο ενό ψηφίσματο για την ανάκαμψη με άφθονε θέσει απασχόληση, σε θέμα για το οποίο θα μιλήσαμε μόλι με την Γενική Γραμματέα τη ΕΤΙΓΙΟΣΥ και για το οποίο ο, πρόεδρος, ο Επίτροπο Αντόρο μα παρουσιάζει ε, τα βασικά στοιχεία. Για τις προφορικές τροπολογίες, ε, τέσσερι τροπολογίες κατατέθηκαν και η κυριαρχική μου πρόταση θα ήταν να φτιάξουμε μια, μάλλον να προτείνω στην ομάδα του ΕΛΚ η τροπολογία 2 να εξεταστεί από την τρίτη γραμμή και μετά ως μια επιπλέον ερώτηση. Έτσι δηλαδή η προφορική ερώτηση θα, περιέχει τέσσερα σκέλη στην ουσία και το κείμενο θα λέει τι συγκεκριμένα σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν μέχρι το τέλος του κειμένου. Αυτό το κομμάτι δηλαδή θα είναι το τέταρτο σκέλος, μια ερώτηση συγκεκριμένη. Για την τροπολογία 1 του ΕΛΚΑ θα πρέπει να πω ότι δεν είμαι υπέρ γιατί πιστεύω πως η κατάσταση της απασχόλησης έχει υποβαθμιστεί σε πολλά κράτη-μέλη Νομίζω ότι το αρχικό κείμενο είναι πιο ε, κοντά στην πραγματικότητα. Τροπολογία 3. Pense qu'on peut euh, le, le, la deuxième partie euh, est intéressante. J'ai plus de problèmes. Το δεύτερο τμήμα είναι πιο ενδιαφέρον, ενώ το πρώτο είναι πιο προβληματικό. Και η τροπολογία 4. Μου φαίνεται κάπως προκατελημένη σε σχέση με το θέμα που προτείνουμε. Όχι, την 4 μπορούμε να την υποστηρίξουμε, νομίζω. Voilà, sur le texte de la question orale, est-ce qu'il y a des... Για το κείμενο της προφορικής ερώτησης υπάρχουν ερωτήσεις ευκρινήσεις. Η κυρία λοιπόν, Μοχά. Α, δεν μου είχατε ζητήσει το λόγο. Τηλεφωνάτε κιόλα. Μάστε. Ο κύριο Όρη. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα τι νόημα έχει μια ξεχωριστή ερώτηση με βάση την τροπολογία 2. Γιατί είναι απαραίτητη αυτή. Είναι απαραίτητη γιατί αν θέλετε γιατί το πρώτο ερώτημα αφορούσε τα διακυβευόμενα σε σχέση με τους μισθούς, τις αποδοχές. Ενώ τώρα που έχουμε τροποποιήσει αυτή την ερώτηση δεν θέτει το θέμα των αποδοχών αλλά του επίπεδου ανεργίας. Είναι πολύ διαφορετική ερώτηση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ζητήσουμε ότι η Κομισιόν μας πει και για το επίπεδο το μισθολογικό, δηλαδή την ε, <clears throat> πολιτική ανάκαμψης μέσω της ζήτησης και επίσης να την εγκαλέσουμε γενικότερα όπως ζητήσατε σε σχέση με την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιότερα των νέων και της χρήσης των διαρθρωτικών πόρων προς την κατεύθυνση αυτήν. Si vous voulez, on peut en reparler. Euh, euh, και euh, θέλετε, μπορούμε να Και d'autres commentaires là-dessus. Εκτός αν υπάρχουν άλλα σχόλια. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό σήμερα, κύριε Ωρί. Εγώ θα προτιμούσα να επαναληφθήσω. Alors, sur euh, les autres propositions de... 73 είναι οι τροπολογίες ε, για τις οποίες έχετε λάβει 11 συμβιβαστικές, ε, τις οποίες συνέταξα εγώ. Βάσει όμως ε, σύνταξης που προετοίμασε η Γενική Γραμματεία γιατί ε, πρέπει να κάνω συμβιβαστικές τροπολογίες ε, επί, βάσει τροπολογιών ε, τις οποίες δεν έχω συντάξει εγώ η ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει για τις τροπολογίες 2, 3, 4 η βασική ήταν η τροπολογία των φιλελευθέρων που λέει διαγραφή την αναφορά στο επίπεδο της, απασχο... της, αναφορής... της αναφοράς στο επίπεδο της απασχόλησης και προσαρμογή με αίτημα της ομάδας ECR για να ληφθεί υπόψη η διαρθρωτική αδυναμία, κάτι το οποίο το έχουμε ενσωματώσει ε, στην ε, συμβιβαστική τροπολογία. Υποθέτω ότι θα το διαβάσατε. Δεύτερη συμβιβαστική τροπολογία αφορά τις τροπολογίες 20 και 21. Δεν νομίζω να δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα οι τροπολογίες αυτές ε, ε, και η τρίτη συμβιβαστική τροπολογία αφορά τις τροπολογίες από 26 έως 29. από όλες τις ομάδες εκτός των σοσιαλιστών και αφορά το θέμα της ε, φορολόγησης ε, της εργασίας και της μεταφοράς του βάρους αυτού ε, και μετά πάμε στην τροπολογία 4 τη συμβιβαστική που καλύπτει τις 38 και 39 και αναφέρει την καταγγελία ε, των ε, καρνητικών συνεπειών. Έχουμε και τη συμβαστική τροπολογία ε και αν θέλετε να κάνουμε και μια συζήτηση για να μπορέσουμε αύριο να ψηφίσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε, στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα ήθελα ευθύ αμέσω να σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις, μια στρατηγική κατάλληλη για ε, ε, και βιώσιμες συντάξεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι όλες ιδιαίτερως που έχω τη δυνατότητα σήμερα να παρίσταμε εδώ και να σας παρουσιάσω σύντομα τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις και επίσης βέβαια να ακούσω και κάποιες ερωτήσεις στο τέλος την αρχή των εργασιών ε, για την ανάπτυξη της επίσημης ε, τοποθέτησης του Κοινοβουλίου για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, δημοσίευσε τη Λευκή Βίπλο ε, μία, ένα, πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για βέβαιες και βιώσιμες συντάξεις στις 16 Φεβρουαρίου για να μπορέσουμε να, μπορέ, να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις του, των συντάξεων και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκές ε, εισόδημα ε, στους ε, συμπολίτε μας μετά τη σύνταξή του, μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ε, δεν χρειάζεται να σας πω για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικές οι συντάξεις, ποιες προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι επηρέασε τη Λευκή Βίβλο. Ε, σήμερα οι συντάξει ε, είναι το ε, βασικό εισόδημα του ενός τετάρτου των συμπολιτών μας και οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει επίσης να μπορούν να βασίζονται στις συντάξει τους κάποια στιγμή και ελπίζουμε να υποβελούνται όχι μόνο από βασική προστασία κατά της φτώχειας αλλά ελπίζουν να έχουν και ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής μετά τη συνταξιδότησή τους. Αλλά αυτό βέβαια ε, σημαίνει και ένα τίμημα. 11,3% του ΑΕΠ από τους δημόσιους προπολογισμούς δαπανήθηκε για τις ε, συντάξεις. Ε, περίπου 13% του ΑΕΠ θα είναι μέχρι το 2016 σύμφωνα με την έκθεση για τη γύρανση που μόλις δημοσιεύθηκε του 2012. Όσον λαμβάνονται βέβαια υπόψη το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και το, ε, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ε, το ενεργητικό ε, δυναμικό μειώνεται σιγά σιγά καθώς η γενιά του baby boom πλησιάζει προς τη συνταξιοδότηση με 6 εκατομμύρια λιγότερους ε, ε, συμπολίτες μας στο ενεργό δυναμικό. Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο δημοσιονομικό αντίκτυπο ε, της γύρανσης. Όλο και περισσότερο βασιζόμαστε ε, σε ανθρώπους ε, ε, που όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο βασιζόμαστε σε ανθρώπους που βρίσκονται στην παραγωγική περίοδο της ζωής τους. Κάτι το οποίο που σημαίνει για μας ότι πρέπει να περάσουμε σε μία μεταρρύθμιση. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης κατέστη σημαντικότερη λόγω του αντικτύπου της κρίσης και στην απασχόληση αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Οι συντάξει είναι σημαντικέ όχι μόνο για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση, αλλά και λόγω του αντικτύπου που μπορούν να έχουν στις δημόσιες δαπάνες και στις χρηματοοικονομικές αγορές. Οι συντάξει ε, είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο αποφασίζουν κυρίως τα κράτη-μέλη, όλο και περισσότερο όμως αποτελούν αντικείμενο κοινή ανησυχία στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο της. Βάσει αυτών των στοιχείων ε, δημοσιεύσαμε για το θέμα αυτό μια πράσινη βίβλο τον Ιούλιο του 2010. Ε, το έγγραφο αυτό δρομολόγησε μια συζήτηση για το πώς το ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να, υποστηριχθεί, να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη στην εξασφάλιση κατάλληλων και παρκών συντάξεων για τους Ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη ε, του χρόνου εργασίας, των ε, ετών εργασίας, ε, της ηλικία συνταξιοδότησης και ε, άλλων τέτοιων παραγόντων. Ήταν ιδιαίτερα έντονη διαβούλευση. Λάβαμε υπόψη μας και την επίσημη τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λάβαμε στοιχεία από πολλές επιτροπές, μεταξύ των οποίων βεβαίως και από τη δική σας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα να ήταν λοιπόν μια ευρύτερη ε, προσέγγιση ε, την οποία ακολουθήσαμε για το συγκεκριμένο ε, έγγραφο. Λάβαμε υπόψη οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια αγοράς και βέβαια αναγνωρίσαμε και τις συνεργασίες αλλά και το όφελος που μπορεί να προκύψει. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν ότι πρέπει να ενισχύσουμε μια αποτελεσματική ε, συνταξιοδοτική περίοδο. Ε, αυτό σημαίνει βέβαια αναμόρφωση και ε, της, του επαγγελματικού βίου, ενίσχυση των προϋπολογισμών για τις συντάξεις. Το 2011 σε 16 χώρες μέλης υπήρξαν συστάσεις συγκεκριμένα για τις, ε, ε, για τις συντάξεις ε, και σε πέντε από τις χώρες αυτές αναφερόταν το ζήτημα σε σχετικά μνημόνια συνεννόησης. Στη συνέχεια το 2012 ευθυγραμμίστηκαν ε, ε, τα στοιχεία αυτά με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ε, με την πρώιμη συνταξιοδότηση, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως επίσης και τη συμπληρωματική, τα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση του εισοδήματός τους μετά τη συνταξιοδότηση. Έχουμε σήμερα τα σχετικά στοιχεία και βλέπουμε ότι οι συντάξει ε, σε 17 ε, κράτη-μέλη ε, εξακολουθούν να είναι αντικείμενο συστάσεων. Βασιστήκαμε λοιπόν σε όλη αυτή τη δουλειά, στην Πράσινη Βίβλο, στη διαβούλευση, όπως επίσης και στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, όπως επίσης και τις συστάσεις για τις διάφορες χώρε Και η Λευκή Βίβλο τονίζει ιδιαίτερα ότι παρά τις προκλήσεις ε, του γυράσκοντος πληθυσμού μπορούν να παραμείνουν επαρκείς οι συντάξεις αρκεί να αναλυφθεί δράση τώρα. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ε, εξασφάλιση μεταξύ του χρόνου ε, του επαγγελματικού βίου και του συνταξιδοτικού χρόνου λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ε, βέβαια, το να αυξηθεί το ηλικιακό όριο σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη ναι, η μακροβιότητα. Ε, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει βέβαια και τη βιωσιμότητα του προγράμματος της σύνταξης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ε, μία αύξηση των συνταξιδοτικών ε, δικαιωμάτων ε, βάσει της καλύτερης ασφάλειας στον χώρο της υγείας και της προσαρμογής των χώρων εργασίας, της ανάγκες όλων των εργαζομένων. Να δώσουμε ευκαιρίες για προοδευτική συνταξιοδότηση και να αλλάξουμε τη στάση των εργαζομένων για να δούμε κατά πόσο η συνταξιδοτική ηλικία που προβλέπεται για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους είναι η κατάλληλη ή όχι. Ε, λήφθη επίσης υπόψη το γεγονός ε, ότι είναι διαφορετική η δυνατότητα συνταξιοδότησης ε, στα διάφορα κράτη-μέλη, 60 ε, ή 65 ανάλογα με τι χώρες, ε, και ότι η πρώιμη συνταξιοδότηση συμβαίνει κυρίως στις χειρονακτικές εργασίες. Επίσης, προσπαθούμε να διευκολύνουμε ε, τους Ευρωπαίους πολίτες να παραμένουν στο ενεργό δυναμικό ε, όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν, ε, δυνατότητα, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ όσων δουλεύουν και όσους δεν δουλεύουν προκειμένου να τους βοηθήσουμε να συμμετέχουν στην αγορά ε, εργασίας και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολλές πολιτικές ε, ε, υποστήριξη κυρίως των γυναικών για να μπορέσουν να συγκεράσουν τον, ε, τις, ε, τις, τον τις οικογενειακές τους ανάγκες με τις επαγγελματικές, ε, οι νέοι να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Επίσης, να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία να δουλέψουν στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει βέβαια ε, ότι το όφελος από ε, χαμηλότερε συντάξει μπορεί να αντισταθμιστεί από το γεγονό ότι κάποια άτομα θα παρημένουν στην αγορά, εργασία, εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η, Λευκό, η Λευκή Βίβλο αναφέρει μέτρα ενίσχυσης τη αποτελεσματικότητα. ε, ε μέσω μιας κινητικότητας, ε, για παράδειγμα, γιατί συχνά χάνουν σε συμπληρωματική ε, σύνταξη όταν πηγαίνουν από τη μία χώρα στην ε, άλλη. Το 2005 προτείναμε μια οδηγία για την, το δυνατό, τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. οι απαντήσει στην Πράσινη Βίβλο έδειξαν ε, ότι χρειάζονταν, χρειαζόταν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ε, για την διατήρηση του συνταξιδοτικού δικαιώματος, αλλά ε, να δώσουμε λιγότερη έμφαση στη δυνατότητα μεταφοράς. Ως εκ τούτου θα ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν έχει κάνει σαφές μέσα στην πράξη για την ενιαία αγορά ότι είναι προσιλωμένη στο να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό το 2012. Θα συζητήσουμε και με την Κυπριακή Προεδρία, την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία, για να ε, προσπαθήσουμε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο πριν από το τέλος του έτους. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι το θέμα του φύλου. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να είναι φτωχές όταν ε, παίρνουν σύνταξη από ότι οι άνδρες και πρέπει να δούμε τη διάσταση του φύλου. Γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά συνήθως συνταξιδόνται νωρίτερα από τους άνδρες και καλύπτονται πολύ πιο σπάνια από συμπληρωματικές ε, συντάξεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αυτό επηρεάζει την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί στην λευκή μας βίβλο είναι και ένα παράδειγμα της επιτυχίας της διαβούλευσής μας, όπου το Κοινοβούλιο και ορισμένοι εμπλεκόμενοι είχαν θεωρήσει ότι αυτό το θέμα δεν είχε αντιμετωπιστεί επαρκώς. Πάντα θα υπάρχουν περισσότερα να πράξουμε και πιστεύω ότι <clears throat> με την γνωμοδότησή σας για τη Λευκή Βίβλο το κατανοείτε αυτό ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Το επόμενο βήμα θα είναι να εφαρμόσουμε τα 20 μέτρα της Λευκής Βίβλου σε συνεργασία και εταιρική σχέση μαζί με τους εμπλεκόμενους. Είναι απαραίτητο να έχουμε πάντα μαζί μας όλους τους εμπλεκομένους. Θέλουμε να έχουμε μια πραγματιστική προσέγγιση και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε οι συντάξει να είναι και να παραμείνουν επαρκείς και βιώσιμες. Ένα από τα πρώτα στοιχεία που περιλαμβάνει ως αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν το, η Λευκή Βίβλος είναι και οι προτάσεις οι οποίες εκπονούνται μαζί με την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων και θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Οικονομικών Θεμάτων στις 21 Ιουνίου και θα είναι το συμπλήρωμα στην έκθεση για την γύρωση ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί και την επάρκεια και την βιωσιμότητα των συντάξεων. Ο στόχος μας είναι να, έχουμε αρκετά, να έχουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν οι συνταξιούχοι ακόμα και σε μια γυράσκουσα κοινωνία. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, το τονίζει και η Λευκή Βίβλο και ελπίζουμε ότι και η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει την θέση αυτή που έχουμε προτείνει. <clears throat> Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ επίση και για το γεγονό ότι σχολιάσατε την πρότασή μας, τη δική μας θέση του Κοινοβουλίου, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη συζητήσει για την Πράσινη Βίβλο και έχει εκφράσει τις απόψεις του. Ξέρουμε ότι δεν θα δεχτείτε όλα τα, τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, αλλά είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το θέμα της μεταφερσιμότητος των συντάξεων που αναφέραμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο εισηγητές μας. Έχουμε την κυρία Όιμεν Ρόιτεν που είναι η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά έχουμε και τον εισηγητή της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής που θα λάβει το λόγο στη συνέχεια. Κυρία Όιμεν Ρόιτεν. Σας ευχαριστώ κύριε Άντορ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι η Λευκή Βίβλος ε, αντικατοπτρίζει με τρόπο αρκετά πλήρη τις συνέπειες της απραξίας, της αδρανίας μας και επίσης τα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από μια καλύτερη δράση από τη δική μας πλευρά. Αν θέλουμε να έχουν βιώσιμες συντάξεις οι συμπολίτε μας όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον θα πρέπει να δράσουμε και υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Η Κομισιόν το έχει πει σαφώς ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ηλικία συνταξιοδότηση. Λόγω της γύρανσης του πληθυσμού θα απαιτούνται εισφορές επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από τη συνταξιοδότηση. Βλέποντας τώρα όμως το έγγραφό σα, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιε διαφορέ απόψεων. Τι μας λέει η Κομισιόν. Μας δείχνει αυτό τον ωραίο πίνακα για τα κράτη-μέλη και τον εργό πληθυσμό μέχρι τα 64. Στη Σουηδία είναι 17% αυτοί που εργάζονται μέχρι τα 64. Και στη δική μου χώρα 53% εργάζονται ακόμα μετά τα 64. και στο Βέλγιο ακόμα λιγότερο. Επομένως, πέραν της ηλικία ταξιοδότησης που αναφέρθηκε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός το ποσοστό των ανθρώπων που θα έχουν εργασία εφόσον το επιθυμούν μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει και μια μεγαλύτερη ε, βοήθεια από τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλω να υπάρξει αύξηση της ηλικία συνταξιδότηση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις άλλες πτυχές μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 είναι κάπως διαφορετική η διατύπωση. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την αντίδρασή σας σε σχέση με το σημείο αυτό και ένα άλλο σημείο που έχει κάπως κριτικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας στο εξή σημείο. Η εφαρμογή των κριτηρίων φερεγγιότητος για τις ε, συνταξιδοτικά ταμεία σημαίνουν ότι θα πρέπει τα συνταξιοδοτικά ταμεία να έχουν υψηλότερες κεφαλαιοχικές ε, ε, απαιτήσει. Εγώ επειδή είχα ασχοληθεί με τα συνταξιοδοτικά αυτά θέματα, περιμένω να έχω ως ε, εργαζόμενο στο παρελθόν ένα καλό αποτέλεσμα από τις επενδύσεις που έχω κάνει σε σε συνταξιοδοτικό, κεφάλαιο. Είμαι λοιπόν εναντίον υψηλών κεφαλογικών απαιτήσεων στα συνταξιοδοτικά ταμεία, γιατί βλέπουμε σε πάρα πολλά κράτη ότι το αποτέλεσμα αυτών των απαιτήσεων είναι να μειώνονται οι αποδόσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων το έχω πει στον κύριο Μπαρνιέ, ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεν κεφαλογικές απαιτήσει, αλλά όχι τόσο υψηλές που να δημιουργήσουν προβλήματα στους εργαζόμενους. Ένα τρίτο σημείο που έχει να κάνει με την δυνατότητα μεταφοράς των ε, συντάξεων. Στατηγική του 2020 έχει μεγαλύτερη ευελιξία, σαν στόχο, μεγαλύτερη κινητικότητα. Όταν όμως κάποιος αναφέρει το θέμα των συντάξεων, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συντάξει αυτές δεν θα χάνονται όταν μετακινείται κανείς. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η Κομισιόν έχει με τις μελέτες τις οποίες έχει διενεργήσει εξασφαλίσει κατά πόσον μπορεί αυτή η μεταφεσιμότητα των συντάξεων μπορεί να εξασφαλιστεί. Ε, ε, ο κύριος Τόμας Μαν. Πάνω από τέσσερα λεπτά μίλησε η κυρία Όιμερ Ρόιτεν. Σας παρακαλώ κύριε Μαν να είσαστε λίγο πιο σύντομοι. <clears throat> Για τους άλλους δύο λεπτά. Γιατί έχουμε δέκα ομιλητές. Και ο κύριος Τόμας Μαν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εν συντομία έχουμε την παρουσίαση του κυρίου Άντορ αλλά και ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος Ρεν έχουν παρουσιάσει την ε, ε, πράσινη βίβλο. Και αυτό δείχνει τη σημασία που της αποδίδει η Κομισιόν. Υπάρχουν ε, στην πράσινη βίβλο τα πρώτα ερωτήματα και στη λευκή βίβλο οι πρώτες απαντήσεις, οι πρώτες κατευθύνσεις. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το θέμα της βιωσιμότητας των συντάξεων, αλλά όπως λέμε και στα γερμανικά, υποκρύπτεται μεταξύ των λεπτομεριών ο διάβολος. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτές τις βιώσιμες ε, συντάξεις. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με το θέμα της εξασφάλισης της φερεγγιότητος στη συντάξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι οργανώνονται εθελοντικά για να έχουν ένα συνταξιοδοτικό ταμείο. Τι θα γίνει με αυτούς, γιατί τους επιβάλλεται τώρα ένα τόσο υψηλό επίπεδο ιδίου κεφαλαίου που θα πρέπει να έχει το ταμείο τους που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. <clears throat> Τον Απρίλιο του 2011 υπήρξανε ε, ουσιαστικά, υπήρξε ουσιαστικά μια εξέγερση των ε, εργαζομένων και των ε, επιχειρηματιών ακόμα που είπαν κάτω τα χέρια από τα συνταξιοδοτικά μας ταμεία με το Solvency 2 δεν, μπορείτε να, δεν μπορούν να είναι βιώσιμα τα συστήματα αυτά. Κάτι το οποίο <clears throat> ήταν επιτυχές σε κράτη-μέλη, τώρα γίνεται κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή η Ευρώπη καταστρέφει τα επιτεύγματα των κρατών μελών. Και όταν μιλάμε για stress test για άλλες επιχειρήσεις, ασφάλειες και τράπεζες, βλέπουμε ότι υπήρξαν πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν περάσει τα stress test με μεγάλη επιτυχία. Και τώρα, επίσης για το θέμα της μεταφοράς των συντάξεων. Ποια είναι η δική σας θέση μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν Θα θέλαμε όλοι τα χρήματα τα οποία έχουν αποκτηθεί σε μία χώρα να μπορούν να μεταφερθούν σε κάποια άλλη. Θα πρέπει να ξέρουμε και ποιε είναι οι προθεσμίε για να γίνει αυτή η μεταφορά. Αυτό αφορά και τη δική μα επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόληση, αλλά επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή, όπου εγώ είμαι συντάκτη για αυτή την αντίστοιχη έκθεση. <clears throat> αλλά θα πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν με το solvency έχουμε καταφέρει στις χώρες όπου υπάρχουν εθελοντικά συστήματα συνταξιώδης ξεπεράσει όλα τα stress test για το solvency. Δεν σας είπα σε εσά δύο λεπτά, αλλά σας ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε για τις πρώτες αυτές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. είναι γεγονός ε, ότι μιλήσατε, σας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και τη δυνατότητα της γενεάς των ε, ηλικιωμένων εργαζομένων να παραμένουν στην απασχόληση. Όντως υπάρχει και σε αυτό ακόμα μεγάλη ε, διαφοροποίηση. Υπάρχουν χώρες όπου το ποσοστό απασχόλησης είναι σχετικά υψηλό ακόμη και για τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους. Φέτος ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γύρανσης ε, και συζητήσαμε πολλές φορές τι πρέπει να γίνει στις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη και στις χώρες που έχουν πολύ καλές επιδόσεις για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι δυνατότητες και να είναι η αγορά εργασίας πιο ε, περιεκτική. και στις χώρες που υπάρχει ψηλό ποσοστό ανεργίας εξακολουθούν ε, να υπάρχουν προβλήματα και σε αυτή την κατηγορία των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων. Η συλλογή και η ανταλλαγή ε, καλών πρακτικών ε, είναι πολύ σημαντική. Πρέπει όλοι οι εταίροι, οι κοινωνικοί εταίροι, οι κυβερνήσει να δεσμευθούν σε διάφορα επίπεδα και στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Απασχόλησης τον Σεπτέμβριο θα ε, συζητηθούν ειδικότερα τα θέματα των ευκαιριών απασχόλησης ε, για τους ηλικιωμένους εργαζομένους. Ε, οπότε, όσον αφορά το θέμα του Solvency 2, καταλαβαίνω ότι είναι ιδιαίτερη η ανησυχία για το θέμα αυτό και όλοι όσοι συμμετείχαν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Λιρέν και ο Μισελ Μπαρνιέ ε, σε, αυτό το, σε αυτές τις συζητήσεις ε, ανησυχούν όλος ιδιαίτερος. Ε, δεν είμαι ο μόνος που ασχολήθηκε με αυτό, αλλά είναι αλήθεια ότι οτιδήποτε αφορά τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες η ευθύνη είναι του Μισελ Μπαρνιέ. Έγινε και μία ε, διάσκεψη το Μάρτιο στο Βερολίνο που ε, αφορούσε ειδικότερα αυτό το θέμα, ε, στο οποίο βέβαια ήρθα σε επαφή με τον Μισελ Μπαρνιέ και του είπα τις ανησυχίες τις δικές μου. Η άποψη της ε, ΑΕΟΠΑ ζητήθηκε προκειμένου να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Βέβαια δεν είναι δυνατόν απλώς να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε νομοθεσία που υπάρχει ε, σε άλλους τομείς, ε, σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς και να τις αντιγράψουμε απλώς στο θέμα της σύνταξης γιατί τότε η Επιτροπή δεν θα κάνει τη δουλειά της. Κάτι τέτοιο θα τη σταθερότητα ε, συστημάτων ε, σύνταξης που ε, λειτουργούν μια χαρά. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ε, νομοθετική, ειδικότερα όταν υπάρχει ιδιαίτερος, ε, ιδιαίτερη ε, αστάθεια στον τομέα των συνταξιδοτικών ταμείων σε πολλές χώρες. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την αίσθηση της ασφάλειας για τις δημόσιες συντάξεις, για τους συμπολίτες μας, αλλά πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε αυτή την περίπτωση η γάμα δέλτα μάρκτ ε, θα προβεί στις απαραίτητες προτάσεις. Εμείς τουλάχιστον είμαστε ε, απολύτως ανοιχτοί ε, να έρθουμε σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους. Η κοινωνική ευθύνη είναι δική δική μου, δικής μου αρμοδιότητος, είναι κάτι που αναφέρεται και στη Λευκή Βίβλο αλλά και σε άλλα έγγραφα. Έχουμε αρχίσει διαβουλεύσεις ε, με την επερχόμενη Προεδρία, όπως ε, είπα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δούμε πού αλλάζει η ισορροπία στο Συμβούλιο. Όταν ε, πήγα στο Βερολίνο στη διάσκεψη μίλησα και με την κυβέρνηση εκεί και είχαμε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση ε, με το αρμόδιο Υπουργείο. Ε, προσπαθήσαν να τονίσω ειδικέ συγκεκριμένε πτυχέ, όπω επίση και τη νομική βάση που έχει αλλάξει από τον τελευταίο γύρο συζητήσεων. Κάτι το οποίο ε, πρέπει να μην μα διαφεύγει επίση. Αυτό που θέλω να πω όμω δεν είναι και τόσο η νομική πτυχή που πιστεύω ότι καλή είναι και αυτή να την αναφέρουμε. Το θέμα είναι ότι μετά την κρίση θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση της ανάγκης ε, μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, που σημαίνει μεγαλύτερη κινητικότητα. Χώρες όπως η Γερμανία ενδιαφέρονται για την ε, ενθάρρυνση της κινητικότητας ε, των εργαζομένων και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν θα χάνονται αν πάει κάποιο Ποιο για 3-4 χρόνια να δουλέψει κάπου αλλού και μετά πάει σε ένα άλλο κράτος μέλος ε, και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν θέλουμε όλοι να δουλέψουμε από αυτού προ όφελο ολόκληρη ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε κάτι σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να τις προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Άνε ναι, και μία ακόμη ερώτηση τελευταία της κυρίας Όμεν Ράιτεν για την ηλικία συνταξιοδότησης. Ναι, υπάρχει μία ιδέα ε, μεταρρύθμισης. Δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, θα σας ενημερώσω όμως για, όμως για τις ε, περαιτέρω εξελίξεις, γιατί το βασικό θέμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της μεταφοράς των δικαιωμάτων. Το θέμα είναι κατά πόσο το 883 θα μπορούσε να είναι ένα μέσο, γι' αυτό ακριβώς που μας λέτε, για την ε, μεταφορά των ε, δικαιωμάτων. Πρέπει να σας πω ότι είναι αλληλεπικαλυπτόμενες οι συζητήσεις για το θέμα αυτό. Ε, δύο είναι ε, οι φάκελοι, αλλά δεν έχω τίποτε συγκεκριμένο να σας πω από αυτό. Θα σας ενημερώσω όμως. Φρεντερίκ Νταρντέν και μετά η κυρία Μίσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, καταρχήν ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε και έπειτα είπατε ότι αυτό το λευκό βιβλίο στην ουσία και είναι οι απαντήσεις που λάβατε μέσα στο πλαίσιο του πράσινου βιβλίου και είναι αλήθεια ότι βρίσκουμε μια σειρά από θέματα που έχουμε ήδη αναφέρει εδώ και συζητήσει εδώ και η Πρόεδρος σα ανέφερε. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτό το λευκό βιβλίο στην ουσία χαρακτηρίζεται από ένα κάποιο ιδεολογικό προσανατολισμό, όπου στην ουσία περνάμε ε, ως λύση τις ε, επικουρικές συντάξεις και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Σε αυτά τα δύο βασικά στοιχεία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και επιμένουμε σε αυτά. Άρα λοιπόν αυτό απομακρύνεται από την ισορροπημένη έκθεση που είχε φτάσει το Κοινοβούλιο στην έκθεση του για το πράσινο βιβλίο. Αυτή την ισορροπία λοιπόν ε, δεν την βρίσκουμε εδώ σε αυτό το πράσινο βιβλίο. Γι' αυτό και θα επανέλθω σε δύο στοιχεία το ενολική συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να θέλουμε εκ πάση της να αυξήσουμε το ηλικιακό όριο δεξιδότησης θα πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά απασχόληση σε όλες τις ε, ε, ηλικιακές τάξεις ε, και πρώτα πρέπει να προσεγγιστεί η πραγματική ηλικία από την νόμιμη ηλικία από την ηλικία ενηλικίωσης Νομίζω πως αυτό είναι ε, ο πρώτος πυλώνας, ο πιο σίγουρος. Τα ποσοστά απασχόληση. οι άλλοι πυλώνε είναι ενδιαφέροντε, μπορούν να συμπληρώσουν. Αλλά κυρίως θα πρέπει αυτός ο πυλώνας να ενισχυθεί για... και αυτό δεν ακούγεται καθόλου στα όσα λέτε, ούτε στα έγγραφά σα. Δεν υπάρχουν κάποιες συνταγέ ή προτάσεις ε, για νέα φορολογικά, ε, δημοσιονομικά έσοδα, ώστε να στηριχθεί αυτό ο πρώτο πυλώνας. Μιλάτε για την ανάγκη να προχωρήσουμε προς τον τρίτο πυλώνα, αλλά μήπως διεθούν δημόσια κίνητρα για τη μετακίνηση προς αυτό τον τρίτο πυλώνα και έτσι αποδυναμωθεί σε Αυτά τα δύο θέματα ε, μεταξύ άλλων. Η κυρία Χίρση και μετά Ντεμπάκερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, ισορροπία που διακρεί το <clears throat> τη Λευκή Βίβλο σε σχέση με προηγούμενα από αυτά τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και νομίζω ότι υπάρχει ένας πιο ειλικρινής τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Όταν μιλάμε για συντάξεις δεν πρέπει να κοιτάξουμε μοναχα αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα 50 ή στα 60 αλλά να δούμε και την ηλικία που είναι τώρα 30 ετών, τα άτομα που είναι τώρα 30 ετών, ακόμα και 20. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια καλύτερη ασφάλεια και δυνατότητα σχεδιασμού και κάποια βιωσιμότητα και για τους ανθρώπους που είναι τώρα νέοι. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα της απασχόλησης στα πιο ηλικιωμένα άτομα. Αλλά φυσικά είναι σαφές ότι πρέπει σταδιακά να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότηση. Εδώ δεν πρέπει να δώσουμε απαντήσεις οι οποίες είναι απλώς όμορφες και ωρεοποιημένες αλλά και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στις νέες γενιές κάποια ασφάλεια στο σχεδιασμό λοιπόν. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να μεταφέρονται οι, οι Αν θέλουμε να έχουμε μια γενιά εργαζομένων που είναι πραγματικά ε, κινητικοί και μπορούν να εργάζονται σε πολλά κράτη-μέλη, θα πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια της κινητικότητας και των συντάξεων. Μπορούμε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο να μιλάμε θεωρητικά για μια ευρωπαϊκή αγορά ηλικία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν δεν έχει κανείς <clears throat> τη δυνατότητα όταν φτάνει σε επίπεδο σύνταξης να εκμεταλλεύεται την εργασία του σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να δώσουμε μια σταθερότητα στους εργαζομένους. Έχετε περάσει τα δύο σας λεφτά. Συγγνώμη που είμαι τόσο σκληρή, αλλά υπάρχουν και άλλοι ομιλητές και σχεδόν έχω κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Ντεμπακέρ και μετά κυρία Ρενιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και τον κύριο Άντορ για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα των συντάξεων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους λήπτες αποφάσεων. Είναι απλό αυτό. Δεν έχουμε καταφέρει σε καλές εποχές, εποχές παχαίων αγελάδων, όταν ήταν ακόμα θετικά τα στοιχεία για τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα, δεν έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις. Και ακόμα Πολλά από τα συνταξιδοτικά συστήματα έχουν διαμορφωθεί όταν το προσδόκιμο επιβίωση ήταν 65 χρόνια και όχι 80 όπως είναι τώρα. Από τη δική μου πλευρά λοιπόν, στα δύο λεφτά τα οποία έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να πω ότι πολλά κρατημέλη έχουν αντιμετωπίσει μόνο το σύστημα πρώτου πυλώνα σε ενταξιοδότηση. Αυτό είναι Επαλαιωμένο, Θα πρέπει ο πρώτο πυλώνας να γίνει ένα δίκτυο ασφαλεία, όχι μόνο για αυτού οι οποίοι το χρειάζονται, αλλά και για αυτού που δεν έχουν καμία δυνατότητα να καλυφθούν από το δεύτερο ή τρίτο πυλώνα για τη σύνταξη. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να πείσει τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτή τη μεταρρύθμιση γιατί άλλο είναι να συνιστάτε κάτι και άλλο να πίεσετε. Και επίσης ε, εξηγήσατε ποια είναι η θέση σας για την ηλικία συνταξιοδότηση και αυτά τα θέματα έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. τελευταίο σημείο στα 30 δευτερόλεπτα είναι μια καλύτερη κατανόηση για τα συνταξιοδοτικά. Υπάρχουν σε πολλές χώρες η δυνατότητα να έχει κανείς τα στοιχεία ώστε με ένα κλικ στο ίντερνετ να μπορέσει να υπολογίσει κανείς πόση σύνταξη θα έχει και πόσα θα είναι τα πρόσθετα ε, ωφέλη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να βοηθήσει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τους εργαζόμενους στο θέμα αυτό. Είναι ένα σημαντικό θέμα, γι' αυτό ζητώ σε όλους να μην είναι με ιδεολογικές παροπίδες, να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να είναι βιώσιμο το συνταξιδοτικό μας σύστημα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νιέ και ο κύριος Μπουπάκης μετά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στο ότι το 11,3 του ε, των δημόσιων προϋπολογισμών πηγαίνει για συντάξεις. Αλλά τι γίνεται εδώ με τον τρίτο πυλώνα στην Αυστρία, ξεκινώντας από το 2003, 2004, δηλαδή πριν από κάμια δεκαετία χρόνια, μέσω μιας ε, φιλελεύθερης κατεύθυνσης έχουμε δώσει δυνατότητα φορολογικών ελαφρύνσεων για τέτοιου είδους συστήματα τρίτου πυλώνα. Όλα αυτά όμως δεν αντικατοπτρίζονται στους ε, εθνικούς προϋπολογισμούς. Και υπήρξε μία ασάφεια για τα θέματα αυτά. Ποια ήταν η θέση σας επίσης για την ανάλυση της Λευκής Βίβλου. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλή η ανάλυση της Κομισιόν έχει λάβει υπόψη πολλά στοιχεία και θεωρεί ορθώς ότι ο καθένας <clears throat> θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα, όχι μονάχα οι, συνταξιό, συνταξιούχοι, αλλά και οι άνεργοι και οι νέοι, όλοι αυτοί να έχουν κάποιο δίκτυο ασφαλείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσουν το θέμα της ε, επιβίωσής τους. Εγώ θα ήθελα όπως να ξέρω με ποιο τρόπο θα, εξασφαλίσετε μια συνεκτικότητα σε αυτά τα οποία λέτε. Και μιλήσετε επίσης και για τις γυναίκες και τη σημασία του να δώσετε στις γυναίκες τις κατάλληλες ευκαιρίες. Μήπως είναι κάπως κοινικό αυτό όταν βλέπω μέσα στην χρηματοπιστωτική κρίση που φάνηκε πόσο εύκολα ε, εξαφανίζονται αυτές οι ευκαιρίες για τις γυναίκες και όταν λέτε τώρα στους, ε, στις γυναίκες ότι πρέπει να επενδύσουν σε τόσο ε, αβέβαια συστήματα όπως αυτά του τρίτου, ε, του τρίτου πυλώνα αντί να χρηματοδοτούν τη συντάξη τους ή τα εργαλεία του πρώτου πυλώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πουπάκης και ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Φυσικά χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για, τα κοινωνικά, για κοινωνικά και βιώσιμα συνταξιδικό συστήματα όμως θα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη εφαρμογή τους πέρα από τους όρους ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής και το περιβάλλον, καθώς σε περιπτώσεις αυξημένης ανεργίας και υποαπασχόλησης δεν μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό γιατί ξέρουμε ότι απαιτούνται ικανέ εισφορέ για να εγγυηθούν αυτά τα, οι επαρκέ συντάξει και η βιωσιμότητά του και αυτέ οι επαρκεί εισφορέ υπάρχουν μόνο αν έχουμε αξιοπρεπεί αμοιβέ και θέσει εργασία. Όμω, υπάρχουν περιπτώσει, και εδώ θα ήθελα την άποψή σα, που αυτέ οι μεταρρυθμίσει αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και κοντόφθαλμα, με συνεχείς οριζόντιε περικοπέ που καταργούν κάθε έννοια κοινωνική δικαιοσύνη και ανταποδιωτικότητα που είναι εντελώ απαραίτητη. Όπω επίση, κάποιε περιπτώσει, όπω στην πατρίδα μου, που η μείωση των συντάξεων χρησιμοποιείται για την κάλυψη ελλημάτων του προπολογισμού, οδηγώντα ένα μεγάλο μέρο Ελλήνων συνταξιούχων κάτω από το εθνικό όριο φτώχεια. Τέλος, όσον αφορά τη Λευκή Βίβλο, μπορεί πράγματι να αποτελέσει ένα σοβαρό εργαλείο για την αδιοργάνωση και τη βιωσιμότητα των συνταξιωτικών συστημάτων. Αλλά αρκεί να μην χρησιμοποιηθεί σαν έναν άλοθη για αποφάσεις που θα μετατρέψουν τη σύνταξη σε ένα προνοιακό επίδομα, οδηγώντας τους δικαιούχους της στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό θα ήθελα να ξέρω αν μπορεί να διασφαλιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προτείνω να ξαναδώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. Δεν θα έχει πολύ χρόνο, αλλά... Ε, μετά θα ακούσουμε τους έξι τελευταίους ε, ομιλητές. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποιες που ελπίζω θα θεωρηθούν βασικές. Ας πούμε για τον αυστριακό τρίτο πυλωνό μπορώ να σας πω ότι ήμουν με τον κύριο Γιώργο Φίσερ και εκείνος ηγήθηκε τις όλες προσπάθειες για το πράσινο βιβλίο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, περί τίνος πρόκειται. Τώρα είναι ιδεολογική υπόθεση όχι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ε, να επιμείνουμε στο θέμα της δημογραφικής αλλαγής και μετατροπής της Ευρώπης. Είναι η βασική τάση, πολλά στοιχεία έχουμε εδώ και το θέμα είναι και κάποιος το ανέφερε αυτό, ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν ε, κατάφεραν να λάβουν τα σωστά μέτρα γιατί υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να αναβάλεις για την επόμενη κυβέρνηση. Τώρα όμως έχουμε φτάσει στα όρια σε κάθε χώρα η επόμενη κυβέρνηση έχει αναλάβει. Και αυτό εν μέρει λόγω του ότι οι δημογραφικές αλλαγές έχουν ε, πια σκάσει, έχει μειώσει, μειώνονται οι γεννήσεις, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει λιγότερο εργατικό δυναμικό, μάλλον σε ηλικία για απασχόληση. Και γι' αυτό δεν ε, μ' αρέσουν αυτά που λέγονται ότι πρέπει να αντιστραφούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει παλιότερα σε κάποιες χώρες, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό. Δεν νομίζω πως είναι ιδεολογικό το θέμα, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε έναν χαρακτήρα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια επιλογή όταν ξεκινάμε τέτοια δουλειά. Είτε θα ενσωματώσουμε κάθε λεπτομέρεια που προέρχεται από τη διαβούλευση και, κάθε, και να έχουμε ένα είδος ευχολογίου, ε, ή να διατηρήσουμε τα βασικά μηνύματα και να φτιάξουμε ε, την απαραίτητη επιχειρηματολογία και προτάσεις γύρω από αυτές τις βασικές ιδέες. Αυτή τη δεύτερη ε, επιλογή κάναμε. Γι' αυτό και δεν βλέπετε διάφορα ελκυστικά θέματα ας πούμε, δεν έχουμε τη συζήτηση για το επιδόματα και τις συνεισφορές και τα λοιπά. Αυτό το αφήσαμε απ' έξω. Αν και πολλοί κόσμος θα χαιρόταν με τέτοιου είδους ε, ε, επίμαχα θέματα. Δεν μιλήσαμε για πολιτικά θέματα, για, για τους ιδιωτικούς τομείς, τον τρίτο το υποχρεωτικό πυλώνα, αλλά είπαμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για το σχεδιασμό του συνταξιδοτικού του συστήματος. Αν θέλουν να έχουν μεγαλύτερο ιδιωτικό τομέα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε, μπορούμε να πούμε ποιος θα ήταν ο σωστός, η σωστή προσέγγιση. Πάντως τα κρατημέλη τα ίδια, δηλαδή το σχεδιασμό των πυλώνων και τη σύσταση, θέλουν να διατηρήσουν την εθνική τους αρμοδιότητα και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. But what is... Και τέλος, είναι κοινή συνεννόηση και σαφές για όλους ότι πρέπει να δουλέψουμε για μεγαλύτερη απασχόληση όντως, μεγαλύτερα ποσοστά απασχόληση και δεν πιστεύω πως οι προτάσεις για την ε, υποχρεωτική επικουρική σύνταξη είναι αντιφατική, αντιφατικές αν είχαμε κάποιο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ίσως υπάρχει εδώ παράδοξο ε, ε, σχήμα όταν μιλάμε για ε, χρονικές περιόδους μεγάλης ανεργίας. Αλλά αυτό το έχουμε το σύστημα σχεδιάσει για μακρά περίοδο. Δεν το έχουμε σχεδιάσει μόνο για τώρα που είναι μεγάλη ανεργία. Όντως πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε όλες τις τάξεις τις ηλικιακέ, αλλά αυτό το πακέτο είναι σημαντικό για τους νεότερους, γιατί οι νέοι που αρχίζουν να δουλεύουν τώρα θα πρέπει να ξέρουν ε, ποιο ήταν το σύστημα και πώς αυτό σχεδιάστηκε ε, για όταν θα συνταξιδοτηθούν χρόνια αργότερα. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Και τέλος φυσικά η ελληνική κατάσταση είναι δυσκολότερη. Ε, γιατί είναι ένα παράδειγμα και όχι το μόνο όπου οι μεταρρυθμίσεις που οφείλονται στις δημογραφικές αλλαγές δυστυχώς συνέπεσαν με την ανταπόκριση στην κρίση που απαιτεί τεράστιες δημοσιονομικές προσαρμόγες πράγμα το οποίο δυσχεραίνει και την μεταρρύθμιση της συνταξιδοτική βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η δημοσιονομική προσαρμογή ούτως ή άλλως δεν θα ήταν απαραίτητη. Ε, και βέβαια η δουλειά των Υπουργών και όλων των φορέων εκεί είναι εξαιρετικά σκληρή και δύσκολο να εξηγηθεί καθώς και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, τα σωστότερα μέτρα. Δεν θα ζήλευα καθόλου τον Υπουργό που πρέπει να τα κάνει αυτά. Ο κύριος κύριος Σύρκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν εδώ Το λευκό βιβλίο μα επιτρέπει να είμαστε πιο αντικειμενικοί και νομίζω πω και το επίπεδο ανάλυση είναι πολύ πιο σοβαρό σε σχέση με το προκάτοχο του, δηλαδή με το πράσινο βιβλίο. Βασικά, Τι λέει εδώ το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τα 27 κράτη-μέλη, σύντομα 28, με ένα σωρό διαφορετικά συστήματα. Εσείς, ε, μάλλον, οι δυνατότητες που έχουμε σε ρυθμιστικό επίπεδο είναι σχετικά περιορισμένες όσον αφορά την χρηματοδότηση, ίσω και όσον αφορά τις ε, τον πολιτικό συντονισμό. Αν λοιπόν θέλουμε να δούμε αυτά τα 20 προγράμματα δράσης, θα δούμε ότι το καθένα απαιτεί συγκεκριμένες ε, προσπάθειες και σίγουρα θα πρέπει να τις παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς σκοπεύετε να οργανωθείτε, με ποιο χρονοδιάγραμμα, πώς θα διερθωθεί δηλαδή αυτό το πρόγραμμα δράσης και θα προχωρήσει. Και έπειτα, θα ήθελα επίσης να καταλάβω αν η Κομισιόν θεωρεί απαραίτητο να δημιουργήσει κάποιο είδος ε, υπηρεσία σε κάποιον οργανισμό για να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Ένα είδος ε, κέντρου, σημείου που θα συγκεντρώνει σταθερά όλες αυτές τις πληροφορίες. Είδαμε πόσο μεγάλες προσπάθειες χρειάστηκε η Επιτροπή και πόσος χρόνος χρειάστηκε για να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Όμως δεν νομίζω πως μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η ίδια προσπάθεια και γι' αυτό και μιλώ για ένα τέτοιο είδος δομή σε έναν οργανισμό που να μπορεί να διευκολύνει τη δουλειά της Κομισιόν. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ πάντα εκπλήσωμαι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών ε, συστημάτων για να αντιμετωπίσει προβλήματα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Οι συντάξεις οριμάζουν μέσα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, 15, 20, 30 χρόνια. Και τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν λιτότητα και μειώνουν τα κοινωνικά ωφέλη. Θα θέλαμε λοιπόν να τονίσουμε το πρόβλημα το οποίο προκύπτει με τις προτάσεις της ε, Κομισιόν προς την Ισπανική κυβέρνηση για τις, ε, ε, για τις συντάξεις. Με τις προτάσεις αυτές δεν είναι ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση στην Ισπανία με, το, <clears throat> με τη γύρανση του πληθυσμού ή κάποια άλλη ε, κατάσταση. Αλλά οι συντάξεις δεν έχουν βραχυχρόνιο ε, χαρακτήρα. Έχουμε πάντα πρόβλημα όμως με τους ε, ανέργους και έχουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, 40% που θα μπορούσαν να είναι ενεργοί και είναι χωρίς να εργάζονται. Είναι καταστροφική λοιπόν <clears throat> αυτή η κατάσταση όπου χρησιμοποιείται τις ε, συντάξεις για να αντιμετωπίσετε τα δημόσια οικονομικά. Ενώ δεν φταίνει συντάξει για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρξει μια εξασφάλιση της ε, βιωσιμότητας. Η ασφάλεια πρέπει να είναι ένα στοιχείο του συστήματος. Αλλά δεν βλέπω στη Λευκή Βίβλο το τι θα γίνει με εκατομμύρια Ευρωπαίων που μέσα σε 20 ή 30 χρόνια δεν θα έχουν το δικαίωμα να έχουν σύνταξη, δεν θα έχουν κανένα απόλυτο δικαίωμα ακριβώς επειδή οι συνδίκες πρόσβασης στα συνδεδοξιδοτικά ταμεία έχουν καταστραφεί. Αυτό είναι ένα στοιχείο αβεβαιότητος, πολύ πιο έντονο, πολύ πιο σημαντικό από την ε, ε, απειλή της δημογραφικής ε, καταστροφής που πόσες φορές μας την παρουσιάζει. Κύριε Αράπτη και μετά κύριο Δεμπέκερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τις περισσότερες ερωτήσεις που είχα να κάνω, τις... Uh, uh, je ah, ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, τις περισσότερες ερωτήσεις που είχα να κάνω, κυρία Επίτροπε, τις πήραν άλλοι συνάδελφοι και τις έκαναν. Όμως με τις απαντήσεις σας μου δίνετε ερέθισμα για καινούριε ερωτήσεις. Η ερώτηση λοιπόν που έχω να κάνω είναι η εξής. Είπατε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας συνέπεσε η αναγκαιότητα για δημοσιονομική προσαρμογή με την δημογραφική γύρανση. Και σκέφτομαι εγώ, γιατί κοιτάζω γύρω-γύρω στην Ευρώπη και βλέπω Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Μήπως και εκεί αρχίζει να συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τι σκοπεύετε να κάνετε και στις χώρες αυτές. Αυτό είναι ένα ερώτημα που βασίζεται στη ζωή. Ε, και το δεύτερο και τελευταίο είναι ότι μιλάμε συνεχώς για αξιοπρεπή εργασία. Decent work. Είναι ένα ερώτημα που έθεσα και στην κυρία Σεγκόλ που ήταν πριν από σας εδώ. Και το θέτω, το προσεγγίζω το θέμα αυτό με μια άλλη διάσταση. Μιλάμε για την αξιοπρεπή εργασία, decent work έχουμε στο μυαλό μας το θέμα της αξιοπρεπούς σύνταξης. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε την αξιοπρεπή σύνταξη. Και κάτι ακόμη και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, ζητάμε δουλειά και σκεφτόμαστε δουλειά για, για τα περισσότερο ηλικιαμένα άτομα στο πλαίσιο της ενεργούς γύρανσης. Ε, ζητάμε όμως δουλειά και για τους νέους. Υπάρχει μήπως μελέτη που να δείχνει αν οι θέσεις εργασίας διεκδικούνται και από τις δύο κατηγορίες. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Μπεκέρ και η κυρία Λινκεβιτσιού της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο ξέρουν οι εμπειρογνώμονες εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό το οποίο θα έπρεπε να ξέρουμε και εμείς από την πολιτική. Όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η Λευκή Βίβλος πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ένα θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι είναι αποφασιστικό ότι οι ανάγκες μεταρρύθμισης που τις ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνονται στις χώρες μας μόνο μετά από την πίεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Φυσικά είναι η υπόθεση των κρατών μελών το να εφαρμόσουν τις προτάσεις της Λευκής Βίβλου. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε τη σημασία που έχουν αυτές οι στάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να πω και μια λέξη σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Υπάρχει κάτι που είναι σε εισαγωγικά στην παρουσίασή σας, αλλά είναι κομβικό <clears throat> να βελτιώσετε, να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχολησιμότητας των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι μονάχα μέτρα τα οποία είναι βραχυπρόθεσμα, αλλά μία με μακροχρόνια προσέγγιση και η ανάγκη επίτευξης μεταρρυθμίσεων. Για μένα η λευκή αυτή είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό εργαλείο για να πείσουμε τα κράτη-μέλη μας να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και εγώ νομίζω ότι είναι εύστοχο μέσω αυτή η Λευκή Βίβλος για να βελτιώσουμε την πολιτική μας και ιδίως το αίσθημα ευθύνης εναντί των επερχομένων γενναίων και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων. Ευχαριστώ. Κυρία Λίνκε Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον Επίτροπο. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτη, έχετε δεδομένα για τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, για τα κράτη-μέλη εννοώ, για το κατά πόσο μειώθηκαν οι συντάξεις ή όχι. Εγώ δεν έλαβα τέτοιου είδου δεδομένα. Βέβαια, εσεί λέτε στη Λευκή Βίβλο ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ε, πιέζει τι δημόσιε τις δημόσιες ε, δαπάνε και συνεπώ τι συντάξει. Θα ήθελα να ξέρω ποιε χώρε έχουν μειώσει τι συντάξει του. Δεύτερο ερώτημα. Πρέπει όντω να μειώσουμε το όριο συνταξιοδότηση, ε, το όριο ηλικία συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι δεν είναι δημοφιλέ από πολιτική απόψεω, ε, δεν είναι δημοφιλή μια τέτοια δήλωση, αλλά κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη πάρει την απόφαση αυτή. Εγώ δεν έχω δει πουθενά κατάλογο των κρατών μελών ε, ως προς τα μέτρα διατήρησης των ε, εργαζομένων στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι αυτές οι χώρες που μείωσαν τις συντάξεις τους και πώς έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την απασχόληση των ηλικιωμένων όσον αφορά τώρα τις συστάσεις για τα κράτη-μέλη και ειδικότερα για τη Λιθουανία. Μα ζητήσατε να μειώσουμε να μειώσουμε τα οικονομικά κίνητρα όσων είναι στο όριο σύνταξη ε, να συνεχίσουν να δουλεύουν. Το γνωρίζετε όμως ότι η λιθουανική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, έχει ζητήσει να ε, συνταξιοδοτούνται όλοι στα 65. Πώς είναι δυνατόν να συγκεράσουμε τα δύο. Ο κύριος Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, στην αναζήτηση της ε, για τα συνταξιδοτικά συστήματα. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη πέρασαν από τα πρότυπα κατανομής στα πρότυπα κεφαλοποίησης. Αυτά τα πρότυπα ε, τόνισαν τα προβλήματα των αγορών εργασίας που που μπορεί να θέσουν σε δυσκολία ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Το πρώτο αφορά τις γυναίκες που έχουν τη δέσμευση της μητρότητας σχεδόν σε όλες τις χώρες. Αναλαμβάνουν και τη φροντίδα της οικογένειας και των ανθρώπων που αποτελούν αυτήν και έχουν, υποφέρουν και από ε, μισθολογικές διακρίσεις όπως αυτές που σχολιάσαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ. Τελικά, η εξίσωση της συνταξιδοτικής της ηλικίας συνταξιδότησης ε, σημαίνει πολύ χαμηλότερη σύνταξη από ότι οι γυναίκες, από ότι οι άντρες και επειδή έχουν και πιο μακρύ προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι τελικά μπορεί να καταλήξουν φτωχές. Έπειτα, στο μεταπητικό τομέα, σε ολόκληρη την ε, βιομηχανία υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Δύο άνθρωποι μπορεί να δουλεύουν σε μια χαλιβουργία. Ένας είναι ένας τεχνικός που δουλεύει σε ένα γραφείο με το air condition, ενώ άλλος είναι εργάτης που δουλεύει στην υψηκάμινο. Ε, αν βγουν στη σύνταξη με τον ίδιο αριθμό ε, ε, των εργασίας, είναι προφανές ότι μέσα τους θα υπάρχει μια διαφορά ριζική στη δυνατότητα στο προσδόκιμο ζωής που θα έχουν και να μπορέσουν δηλαδή να έχουν την κατάλληλη σύνταξη. Πώς λοιπόν λαμβάνεται υπόψη η διαφορά της, της φύσης της εργασίας και κυρίως της επιβαρυντικής εργασίας. Έπειτα, οι ατυπικές εργασίες η αγορά εργασία έχει γίνει πιο ευέλικτη, ναι, και υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που δουλεύουν για μια χρονική περίοδο, έπειτα σταματούν και έπειτα ξαναρχίζουν να δουλεύουν. Αυτά τα κενά με τα συστήματα με κεφαλαιοποίηση δεν μετράνε, δεν ανταμείβονται, δεν υπάρχουν. Καλύπτονται, υποτίθεται, με αυτή τη συμπληρωματική ε, επικουρική σύνταξη. Εσείς τι θα κάνετε για να καλύψετε αυτούς τους κοινωνικούς κινδύνους. Για να ξεκινήσω με το ερώτημα για τις αρμοδιότητες μας. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε νομικό επίπεδο εδώ, αλλά τα κράτη-μέλη χαιρετίζουν τη δράση της Κομισιόν, την Πράσινη Βίβλο και τη Λευκή Βίβλο. Κάποια κράτη όπως το Βέλιο έχουν και αυτά αυτή την ε, κατεύθυνση με τις ε, λευκές και πράσινες βίβλους. Πολλές χώρες όμως δεν έχουν τέτοια έγγραφα προβληματισμού. Γι' αυτό νομίζω ότι η ανάλυση της Κομισιόν και τα έγγραφα πολιτικής ήταν ιδιαίτερα καλόδεκτα, <clears throat> ακόμα και αν σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε συμφωνία γιατί δίνουν ακριβώς υλικό για προβληματισμό και διάλογο. <clears throat> Υπάρχουν σαφείς σχέσεις μεταξύ των συντάξεων της εργασιακής αγοράς και, της χρημα... και των χρηματαγορών στην Ευρώπη και υπάρχει και σίγουρα μία νομιμοποίηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Το αν χρειάζεται τώρα να υπάρξει ένας νέος φορέας για τα θέματα αυτά, εγώ ξέρω ότι κάποιοι υπάρχοντες φορείς βρίσκουν τον εαυτό τους σε δυσκολία. Υπάρχει μια διαφυσβήτηση της νομιμοποίησης αυτών των φορέων. Η ίδια η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης είναι και, αυτός και αυτή ένας φορέας. Και με την έκθεση για την γύρωση νομίζω ότι έχουν ήδη παίξει ένα σημαντικό ρόλο και με την ε, συζήτηση με τους εμπλεκομένους σε σχέση με τα συμπεράσματα αυτών των μελετών και με την υποστήριξη των προτάσεών μας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Νομίζω ότι φέτος ένα τμήμα αυτών των συστάσεων έτυχαν ταχείας εφαρμογής, ιδίως σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης. Εγώ δεν μου αρέσει αυτό το τμήμα της συζήτησης όταν μονάχα εστιάζουμε στην ηλικία συνταξιοδότησης. Γιατί εμείς έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης σε όλες τις ομάδες ηλικία και σε όλα τα φύλλα. Πρέπει να είμαστε όμως ειλικρινείς ότι σε πολλές χώρες το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 50% ή λιγότερο και πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα για να αυξηθεί το ποσοστό απασχόληση των γυναικών όχι μόνο στην Νότια Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου είναι ένα σημαντικό θέμα. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχει υποστήριξη για παιδικούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς και για την εξάλληψη άλλων εργαλείων που εμποδίζουν τις γυναίκες από το να γυρίσουν στην αγορά εργασίας, θα, το να υπάρχουν ευκαιρίες για διαβίου ε, εκπαίδευση, στοχευμένες δυνατότητες του επιχειρήν, εργασία μερικής απασχόλησης κτλ. Όλα αυτά όμως που να μας δώσουν δυνατότητα να έχουμε συσσόρευση στοιχείων για την ε, κοινωνική ασφάλιση. Σε πολλές χώρες υπάρχουν οι λεγόμενες μίνι εργασίες, τα mini jobs, όπου ζητάμε να υπάρξει σαφής δράση για να μειωθούν οι πρακτικές αυτές και να ευνοήσουμε πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν και μεγαλύτερη κοινωνική ασφάλιση και συσσόρευση ε, ευκαιριών για σύνταξη, γιατί σε μακροχρόνιο επίπεδο μια τέτοια στρατηγική με μίνι εργασίες, εργασίες του, του ποδαριού δεν είναι ουσιαστικά ναι, ναι, κάτι ναι, το οποίο μπορεί να είναι βιώσιμο. Πρέπει να δείτε λοιπόν την ε, επερχόμενη έκθεση για την ε, επάρκεια των ταμείων γιατί η χρηματοπιστωτική κρίση βέβαια επηρέασε αρνητικά τις ε, συντάξεις. Όλες οι χώρες λοιπόν της ε, Νότια Ευρώπη ε, είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά θα πρέπει εδώ να αγωνιστούμε για τι χώρε αυτέ να έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό απασχόληση. Κάποιες ε, χώρες έχουν θέσει και επιχειρήματα λόγω της κρίσης να μειωθεί η ηλικία σας συνταξιοδότησης. Αν κάνετε τους υπολογισμούς, αυτό δεν είναι αδύνατο να θεωρήσετε ότι με το να μειώσετε την ηλικία συνταξιοδότησης στο τέλος της ημέρας θα φτάσετε σε μια κατάσταση που όλοι θα έχουν μια θέση απασχόληση και μετά μπορείτε πάλι να αυξήσετε την ηλικία συνταξιοδότηση. Εμείς όμως θεωρήσαμε ότι ακόμα και οι χώρες που βρίσκονται στα προγράμματα λιτότητος, οι χώρες που διατρέχουν μία <clears throat> κρίση, θα βγουν κάποια στιγμή από την κρίση και θα περάσουν σε μια αρμονική οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια δεν είναι ο στόχος της Λευκής Βίβλου να ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην ιδέα ότι κάποιες χώρες θα μείνουν στο διηνεκές στην ύφεση θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα βρεθούν λύσεις στα προβλήματα της ε, νομισματικής ένωσης και θα υπάρχει μετά εξισορροπημένη ανάπτυξη. Κάποτε. Κάποτε. Και επί τη βάση αυτή θα πρέπει να εργαστούμε για το να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης που τώρα όταν υπάρχει συνεχής πίεση από τις χρηματαγορές είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα κράτη-μέλη έχουν ελάχιστο περιθώριο ελιγμών για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Ώστε θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για αξιοπρεπή αμοιβή εργασία και αξιοπρεπή συντάξει. Πώ θα το κάνουμε αυτό, θέλουμε να αυξηθεί, όπω σα είπα, το ποσοστό απασχόληση και επίση να έχουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συσσόρευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Όταν συζητούσαμε για την πράσινη βίβλο, ο Νίκολα Βάρφ από το London School of Economics μας εξήγησε με μεγάλη σαφήνεια ποιες είναι οι επιλογές που πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η αύξηση της ηλικία ταξιοδότησης θα είναι η μόνη λύση. Μπορούμε να αυξήσουμε και τις συνεισφορές των εργαζομένων. <clears throat> Κάτι βέβαια που έχει ε, αρνητικό αποτέλεσμα για την ε, ανταγωνιστικότητα Μπορεί επίσης κανείς να δεχτεί και μακροχρόνια χαμηλότερες συντάξεις. Αλλά αυτό φέρνει και τον κίνδυνο της ένδυας σε μεγάλη ηλικία, κάτι το οποίο δεν θέλουμε να γίνει. Έχοντας λοιπόν εξετάσει όλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους στόχους και τις παραμέτρους, καταλήξαμε στα συμπεράσματα της Λευκής Βίβλου και σας ευχαριστώ λοιπόν για το ενδιαφέρον σας και τα σχόλιά σας και προσβλέπω στην ε, έκθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Η ανταλλαγή υπόψη ήταν εξαιρετικά πλούσια για ένα θέμα που κινητοποιεί πολύ τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, σας ζητώ όμως να μην φύγετε γιατί έχουμε ακόμα ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη το οποίο θα συζητήσουμε στα αγγλικά.